Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρωινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Με το σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως, απαλλαγή 2009, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παρουσία του ε, Επιτρόπου Αρμοδίου για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπέθρου, κυρίου ε, Τσόλος. Θα δώσω αμέσως τον λόγο στον κύριο Κρετά, εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Το άρθρο 3 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει ε, ε, παρατηρήσεις για τέσσερα θέματα. Ε, γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, προστασία της υπαίθρου, προστασία των καταναλωτών. 57 δις ευρώ, σχεδόν δηλαδή το μισό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το κύριο συμπέρασμα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι οι πληρωμές αυτές έχουν ένα περιθώριο λάθους που εκεί μένεται μεταξύ 2 και 5% αν βάλουμε αυτό το ποσοστό ε, σφάλματος σε μια ιστορική ε, προοπτική πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά υψηλότερο από το 2008 που ήταν μείον 2%. Στην πραγματικότητα το έτος 2008 είναι αυτό που αποτελεί εξαίρεση διότι πάντοτε το περιθώριο λάθους ήταν πάντα παραπάνω από 2% πλην του έτους 2008 για να εκτιμήσει ε, το ε, σφάλμα, περιθώριο σφάλματος ε, στο, στη διάρκεια του έτους το ελεγκτικό συνέδριο κάνει επιτόπου ελέγχους όσον αφορά τις πληρωμές και επίσης κατηγοριοποιεί τα σφάλματα. Πρώτον, σφάλμα επιλεξιμότητος, εάν δηλαδή δεν είναι επιλέξιμος ο τελικός ωφελούμενος δικαιούχος. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ορισμένες παρατηρήσεις το 2009. Ε, μία ΟΤΑ ε, για ένα στάδιο 300 εκταρίων ε, ε, συγγνώμη, 530 εκταρίων, ε, ενώ δεν είναι το δικαιούχα για οποιαδήποτε επιδότηση γεωργική, διότι δεν επρόκειτο για γεωργική καλλιέργεια, παρόλα αυτά θεωρήθηκε δικαιούχος για μια γεωργική εκμετάλλευση σε μια άλλη χώρα. Είδαμε πλασματικές νομικές δομές βάσει των οποίων γεωργοί είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν χτήματα τα οποία δεν είχε στην ε, κατοχή του και αφετέρου ότι ε, ασκούσαν γεωργική καλλιέργεια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και οι δύο περιπτώσεις ήταν πλασματικές, επομένως δεν ήταν δικαιούχος ο συγκεκριμένος άνθρωπος τρίτη κατηγορία σφαλμάτων, το ποσό στο οποίο ανέρχεται η επιδότηση. Δηλαδή, ο δικαιούχος ζητά περισσότερα από αυτά που πρέπει να πάρει. Σε 12 περιπτώσεις, σε ένα κράτος μέλος, καταβλήθηκαν επιδοτήσεις ανώτερες κατά 20% από αυτές που πραγματικά έπρεπε να δοθούν στους δικαιούχους. Τα δύο τρίτα των σφαλμάτων που διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο ε, αφορούν αυτές τις δύο κατηγορίες λάθους που μόλις ανέφερα. Υπάρχει όμως και μία άλλη κατηγορία σφάλματος ε, την οποία ορίζει ε, το ελληνικό συνέδριο ως μη ποσοστοποιήσιμο σφάλμα. Δηλαδή δεν είναι σε θέση το ελεγκτικό συνέδριο να ποσοστοποιήσει την επίπτωση των σφαλμάτων αυτών στον προϋπολογισμό και επομένως αυτού του είδου τα σφάλματα δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στο ποσοστό σφάλματος. Όμως είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα σφάλματα αυτά έτσι ώστε να γίνει μια γενικότερη εκτίμηση της κατάστασης. Επισύρω την προσοχή σας στο θέμα αυτό, διότι τούτο σημαίνει ότι το προαναφερθέν περιθώριο σφάλματος το οποίο ανέφερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα έτσι ώστε να συνυπολογίσουμε την τρίτη κατηγορία λαθών. Δεύτερο γενικό συμπέρασμα του ελεκτικού συνεδρίου αφορά στο σύστημα διαχείρισης των δαπανών, διοικητικό σύστημα, ε, σύστημα πληροφορικής, σύστημα γεωγραφικής αναγνώρισης των τμήματων ε, και ε, σύστημα αναγνώρισης των δικαιούχων συμπεραίνει το ελεγκτικό συνέδριο ότι τα συστήματα διαχείρισης δεν είναι αποτελεσματικά. Βεβαίως αυτό το δεύτερο συμπέρασμα εν μέρη εξηγεί το πρώτο συμπέρασμα, διότι βεβαίως λόγω των ελήψεων στην διαχείριση προκύπτουν τα σφάλματα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω δύο λόγια, δύο στοιχεία ε, για αυτό το οποίο αναφέρω τώρα από την ε, μία πλευρά το Άιαξ και από την άλλη πλευρά το σύστημα ανάκτησης των αχρεωστήτων καταβληθέντων. Το Άιαξ πρώτα. επανειλημμένα το ελεγκτικό συνέδριο λόγω των διασταυρώσεων που έχει κάνει ε, αποτελεί ένα ε, αποτελεσματικό σύστημα και αυτό αποδεικνύεται και από το μέσο όρο σφάλματος του γεωργικού τομέα. Όμως, οι νέες βάσεις δεδομένων που έχουν περιληφθεί στο σύστημα. Μετά από την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος ε, πληρωμών και του ενιαίου συστήματος πληρωμών ανά επιφάνεια. Ε, νέες παραγωγές όπως ε, η ελεουργία ή ο καπνός στην νέα περίμετρο του ΟΣΔΕ είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν διαπιστώνει ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη γεωγραφική αναγνώριση των εδαφών καθώς επίσης και στην εφαρμογή της βάσης δεδομένων όπου καταγράφονται τα μεμονωμένα δικαιώματα ενιαίου, ενιαίας πληρωμής. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο έχει διαπιστώσει ανεπάρκειες όσον αφορά τον έλεγχο επιτόπου από τους εθνικούς οργανισμούς ε, πληρωμής καθώς επίσης ε, και ε, ανεπάρκειες στους ίδιους ελέγχους από τους εθνικούς φορείς πιστοποίησης. Τρίτο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι η επιστροφή των αχρεωστήτων καταβληθέντων τα υπομνήματα τα οποία έχουν ε, δοθεί έχουν αναπτυχθεί περισσότερο το 2009 σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Όμως η κατάσταση των επιστροφών είναι ακόμα εξαιρετικά ανελειπής και ανεπαρκής και επομένως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα βάσει συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Οι πληρωμές ε, έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές ε, και η αμφισβήτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ε, αφορούν τις εθνικές αρχές. Αναφερόμαστε σε 1,3 δις ευρώ τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2006 ακόμα έπρεπε να επιστροφούν 736 ε, εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το μισό της εκατό, δεν είχαν ακόμα επιστραφεί τρία χρόνια μετά. Από τα 736 εκατομμύρια μονάχα 26, 121 εκατομμύρια είχαν δοθεί, είχαν επιστραφεί από τους τελικούς ε, δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπα 411 είχαν επιστραφεί από το ακράτη, που σημαίνει από τους φορολογούμενους. Τέλος, το ελεκτικό συνέδριο μελέτησε την έκθεση δράσης του Γενικού Γραμματέα για την ε, Γεωργία. Διαπιστώνει ότι η μέθοδη που χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας για επιβεβαίωση των στοιχείων δεν ευθυγραμμίζεται και άρα δεν μπορεί να συγκριθεί με την μέθοδο του ελεγκτικού συνεδρίου. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού ε, ε, Διευθυντού ε, το περιθώριο λάθους βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το 2%. Βασίζεται δε στα στοιχεία των εθνικών μονάδων και υπηρεσιών πληρωμών, των οποίων οι ανεπάρκειες και οι ελλείψεις αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επομένως θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε σαν περιθώριο σφάλματος αυτό που ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση. Το ελεγκτικό συνέδριο επίσης θεωρεί ότι, ότι είναι ακόμα πρώιμη η άρση της ε, επιφύλαξης σχετικά με τον ΟΣΔΕ στην Ελλάδα. Πρέπει να πω, περαίνοντας ότι το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει και αναφέρει μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την αποσαφήνιση των κανόνων, την καλύτερη στοχοθέτηση των δικαιούχων και ε, μια γρηγορότερη επιστροφή των αχρεωστήτων καταβληθέντων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ο Επίτροπος κ. Στιόλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Με χαρά παίρνω το λόγο σήμερα για να μιλήσω για το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου της ετήσιας έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου. Προσδίδω ιδιαίτερη σημασία στην σωστή διαχείριση της κοινή γεωργικής πολιτικής, διότι αυτή η διαχείριση η σωστή θα είναι και το κλειδί για την επιτυχία της πολιτικής στο μέλλον. Με τις προσπάθειες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό σφαλμάτων ε, κυμαίνεται ε, γύρω από το κατόφλι του να χαρακτηριστούν ως ουσιώδη ε, σφάλματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας δείκτης της σωστής διαχείρισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και κάνουμε αυτή τη διαπίστωση βασιζόμενη στο δείγμα του ελεγκτικού συνεδρίου 241 περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και έλεγχοι σε επίπεδο κρατών μελών και έχουμε κάνει και ελέγχους εμείς εσωτερικά ε, στη δική μου υπηρεσία, στην υπηρεσία της οποίας προείσταμε. Ωστόσο, αυτό το κεκτημένο δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα εάν δεν διατηρήσουμε τις προσπάθειές μας. Κάθε χρονιά πρέπει να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες για να έχουμε σωστή διαχείριση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε τη δέσμευση ε, των επίσημων κρατικών αρχών στα κράτη-μέλη. Άλλωστε οι στόχοι μας είναι κοινοί. Και γι' αυτό παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ στην ε, εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο κράτους μέλους. Και όταν ε, αυτό αποδεικνύεται απαραίτητο, επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Κάθε φορά εμείς ε, δείχνουμε κόκκινη κάρτα όταν αυτό είναι απαραίτητο. Είναι κάτι που έχω κάνει στο παρελθόν και δεν θα διστάσω να το ξαναπροτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων κάθε φορά που αυτό θα είναι απαραίτητο. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις προόδους που έχουν σημειωθεί έχουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Αυτό το οποίο ε, ονομάζουμε στα αγγλικά IACS. E Είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου. Αυτό το δείχνουν οι έλεγχοι που έχουμε κάνει επί τόπου στην πλειονότητα των κρατών μαλλών, παρόλο που έχουν σημειωθεί, έχουν φανεί κάποιες αδυναμίες στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα στο παρελθόν. Και κάποιες ανεπάρκειες σε ορισμένα άλλα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και ε, με το σύστημα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων. Υποχρεώσαμε τα κράτη-μέλη να κάνουν εις βάθος ετήσια αξιολόγηση αυτού του συστήματος διαχείρισης των αγροτεμαχίων. Και η αξιολόγηση αυτή θα δείξει τις αδυναμίες. Εάν τις δείξει, τότε υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διορθωτικές δράσεις. Και ε, θα κληθούν οι οργανισμοί πληρωμών να ε, αξιοποιήσουν την ε, εμπειρία άλλων οργανισμών πληρωμών προκειμένου να τους φτάσουν και προκειμένου όλοι να είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι λοιπόν ένα πεδίο πάνω στο οποίο θα δράσουμε και στο μέλλον. Δεύτερο πεδίο είναι το θέμα των ανακτήσεων. Έχουμε υψηλότερο ποσοστό αυτών συγκριτικά με το παρελθόν. Καλύτερο δηλαδή από το ε, ταπεινό 10% που αναφέρεται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στα τέλη του 2009 τα κράτη-μέλη είχαν ε, ανακτήσει το 49% αυτών που έπρεπε για το 2007. Ε, θεσπίσαμε τον κανόνα του 50-50 που λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για τα κράτη-μέλη ώστε να αναλάβουν πιο έντονη δράση στον τομέα αυτό. Τρίτο πεδίο που μας αφορά και με το οποίο θα ασχοληθούμε αντώνας είναι η αξιοπιστία αν θέλετε των κρατών μελών. Ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο των οργανισμών πιστοποίησης. Έτσι ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Για να επιβεβαιώσουμε τα ποσοστά σφαλμάτων, οι οργανισμοί πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν αντιπροσωπευτικό δείγμα των συναλλαγών ε, τις οποίες χειρίζονται οι οργανισμοί πληρωμών είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βεβαίως, το μεγαλύτερο διακύβευμα, αν θέλετε, εκεί που θα δράσουμε περισσότερο είναι το, η ευρύτερη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η απλούστευση θα πρέπει να παραμείνει ε, ε, στο προσκήνιο ώστε να δαπανώνται σωστά τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου και να ανακτώνται, να επιστρέφονται όταν γίνεται ε, κακοδιαχείριση. Κάτι το οποίο έχω επανειλημμένως υπογραμμίσει. Χρειάζονται πιο απλή έλεγχη και χρειάζεται επίσης να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μικρών εκμεταλλεύσεων. Και θα πρέπει να απλουστεύσουμε και το ε, θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης και της ε, τήρησης των περιβαλλοντολογικών όρων. Πολύ συχνά έχει γίνει κριτική και από το ελεγκτικό συνέδριο για όσους λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς να ε, ασκούν επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα. Μιλούμε για τους ενεργούς αγρότες. Και γι' αυτό έχουμε συστήσει μια ομάδα ad hoc των διαφόρων κατατόπους ΟΠΕΚΕΠΕ, Οργανισμών Πληρωμών, ώστε να ε, εξεταστούν οι προτάσεις και να δρομολογηθούν. Η κοινή γεωργική πολιτική έχει πολύ σημαντικό προϋπολογισμό και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να κάνω το παν ώστε να, έχει σωστή, να γίνεται σωστή διαχείριση. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του Ευρωπαίου πολίτη και για να το κάνουμε αυτό πραγματικά χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη στήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία. Ο εισηγητής, κύριος Χατζημαρκάκης. Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Τσόλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση. Βλέπουμε ότι κατέχετε την υπόθεση αυτή καλά, το θέμα αυτό. Είχατε άλλωστε αντίστοιχη ενασχόληση και στην πατρίδα σας στο Υπουργείο ε, Γεωργίας. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλά. Ταυτόχρονα ο κύριος Κρετά επίσης έχει εξαίρετη γνώση της γεωργίας και πριν από την ανάλυση των δραστηριοτήτων στο Ελεκτικό Συνέδριο στη Γαλλία, την πατρίδα του, που έχει πολύ μεγάλη, όπου έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια ο γεωργικός τομέας. Έχουμε να κάνουμε το μεγαλύτερο ε, κεφάλαιο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίες και κύριοι. Οι επικρίσεις ακούγονται, πολλές επικρίσεις που πάντοτε δεν είναι και αιτιολογημένες. επικρίσεις ε, Φερρυπίν για τα συστήματα επαγρύπνησης, παρακολούθησης, ε, τα οποία όμως κατά λειτουργούν. Και βλέπουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φερρυπίν για το σύστημα IAX, ότι υπάρχουν ε, αποκλήσεις σε θέσεις ε, δαπανών, όπως αυτές οι οποίες συστήσαμε χθε, οι οποίες χάρη στο σύστημα IAX αντιμετωπίζονται. και αντιμετωπίζονται παρά το ότι είναι μοιρασμένη η διαχείριση των προγραμμάτων. Πράγμα στο οποίο πάντοτε διατυπώνουν τι ε, επιφυλάξει του οι εκπρόσωποι τη Κομισιόν, ότι δηλαδή όπου υπάρχει μοιρασμένη αρμοδιότητα τα προβλήματα είναι πιο αυξημένα. Βέβαια παραμένουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και κύριε Επίτροπε θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τα συνεχιζόμενα προβλήματα τα σχετικά με την Ελλάδα διότι ξέρουμε ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί και θα ήθελα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι σαφής βέβαια οι επικρίσεις που ακούστηκαν αλλά δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Πολλά έχουν καταφέρει στην εφαρμογή του Άγιαξ, αλλά δεν έχουν λύσει κάθε πρόβλημα στην Ελλάδα. Και έτσι θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε το μέλλον ε, για να ε, ενημερωθούμε για το μέλλον και στη Γεωργία και στην Ήπεθρο ώστε να έχουμε στοιχεία αντίστοιχα με αυτά τα οποία ε, γνωρίζουμε στην πολιτική συνοχής δηλαδή ε, ξέρουμε ότι εφόσον η τωρινή επι... εποπτεία στηρίζεται στις άμεσες πληρωμές θα δυσκολέψει πολύ η εποπτική δουλειά με την εξέλιξη στον τομέα αυτών της γεωργίας, όπως συνέβη και στην συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε σχέση με το ΟΣΔΕ, με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, η Άγιαξ, τι στοιχεία έχετε και τι προτάσεις βελτίωσης μπορείτε να προσφέρετε. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να δούμε πού εντοπίζονται τώρα τα προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τους κανόνες, με τις διατάξεις και με την ερμηνεία αυτών. Και θα ήθελα, αναφερόμενο και προ τι δύο προσωπικέ εδώ πλευρέ, δηλαδή και προ την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ρωτήσω γιατί δεν ακολουθούμε το σύστημα που έχουμε στη συνοχή, δηλαδή τι τριμερεί συνομιλίε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ό,τι φαίνεται στι δειγματοληψίε του, έχει μια σχεδόν αυτόνομη δράση. Στο τρόπο με τον οποίο οι παραδείγματι αντιμετωπίζονται οι πράσινες εκτάσεις, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί δεν υπάρχουν τριμερεί ε, συνομιλίε, γιατί δεν μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση εξηγήσει. Σε τελευταία ανάλυση, οι πράσινε εκτάσει είναι άλλο πράγμα στην... Ε, και είναι άλλο πράγμα και ερμηνεύεται διαφορετικά στη Σκωτία και είναι άλλο πράγμα στη Βουλγαρία, Φερρυπίν. Και ναι δεν υπάρχει ε, ε, ανάγκη για ερμηνεία ιδιαίτερη σε κάθε περίπτωση, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος κατάλογος βασικός των στοιχείων που πρέπει να περιελαμβάνει ο ορισμός κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάτσουν η Επιτροπή, το Ελεκτικό Συνέδριο και οι κυβερνήσεις μαζί στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε κάθε κατηγορία ε, που τους απασχολεί στην πολιτική αυτή για τη γεωργία, τι ορισμούς δίνουν. Όπως, σε παραδείγμα, στην περίπτωση του περίφημου ε, αγρότη του καναπέ της Ιρλανδίας. Τι σημαίνει αυτή η ερμηνεία, τι σημαίνει αυτός ο όρος. Επίσης συγκεκριμένα ε, και για τον κύριο Κρετάν αλλά και για την Επιτροπή γιατί συνεχίζει η Ελλάδα να ε, εισπράττει χρήματα να συνεχίζονται δηλαδή αυτές οι καταβολές ενώ δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην υλοποίηση του συστήματος ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εφόσον το κράτος δεν ε, συμμορφούνται με τις υποχρεώσεις του γιατί εξακολουθεί να εισπράττει χρήματα. Και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε πιο ε, ελαστική. Στην ερώτηση υπαριθμών 16, Φερρυπίν. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά τα πιστοποιητικά και οι εκθέσει, γιατί εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει χρήματα, αυτό βέβαια αφορά διαφορετικά περισσότερα κράτη, και λαμβάνω την εξή απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Έχουμε ένα από καιρό παγιωμένο σύστημα πληρωμών. Λαμβάνουν προκαταβολές τα κράτη-μέλη πληρωμές οι οποίες στη συνέχεια εντός εισαγωγικών νομιμοποιούνται, εντός εισαγωγικών νομιμοποιούνται από το κράτος μέλος με την ε, παραγωγή των ε, ισολογισμών τους που ελέγχονται δημοσιονομικά. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Δηλαδή, προ, προκαταβάλλεται τα ποσά, πολύ καλά, παγιωμένη πρακτική, το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά όταν ένα κράτος μέλος Παγίος παραβιάζει τους κανόνες, όταν ξέρετε ότι παραβιάζει τους κανόνες, πώς είναι δυνατόν να συνεχίζετε τις αυτό Εκείνο που δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν υπάρχουν, Φερρυπίν, μέτρα παραδειγματισμού, γιατί δεν υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα. Όταν ένα κράτος μέλος επανειλημμένο παραβιάζει τους κανόνες, γιατί δεν του, ε, ε, ε, δεν του λέτε ένα λεπτό τα λεφτά αυτά δεν μπορείς να τα πάρεις πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματά η καταβολή των ποσών όταν ξέρουμε ότι ακολουθεί ένα σταθερό, μια σταθερά ένα κράτος και η σταθερά αυτή είναι η παραβίαση των κανόνων. Το είδαμε με την Ελλάδα. Δέκα χρόνια χρειάστηκε για να ε, επιβληθούν ε, οι σχετικές κυρώσεις, μάλλον να αντιληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και εκεί είδαμε όντως μια κάποια βελτίωση. Αλλά μεταξύ είχαν περάσει δέκα χρόνια που πλήρωνε ο Ευρωπαίος και επίση θα επανέλθω σε αυτό το οποίο εδώ και 10 χρόνια οπωσδήποτε έχουν πει οι συνάδελφοι και κυρίω ο κύριο Μιλτερ ο οποίο αγωνίζεται για την υπόθεση αυτή εδώ και χρόνια. Θέλουμε δηλώσει από τι εθνικέ αρχέ. Η δήλωση μια εθνική αρχή είναι ο καλύτερο τρόπο, το καλύτερο εργαλείο που μπορούμε να έχουμε στη θέσή μα για να εξασφαλίσουμε σαφήνεια από τα κράτη-μέλη. Ο Υπουργό Γεωργία τη Ελλάδα που έρχεται εδώ και εκτίθεται ζητώντα χρήματα, θα πρέπει και να είναι υπόλογο σε περίπτωση κακοδιαχείριση. Και αυτή είναι η πρωταρχική μα διεκδίκηση. Δεύτερον, κύριε Τσόλο, είπα και νωρίτερα ότι η έκθεση δραστηριοτήτων υπογράφεται από το Γενικό σα Διευθυντή. Πολύ καλά. Είναι εντάξει, είναι καθαρή έκθεση ε, πλην όμως θα ήθελα να δω και τη δική σας υπογραφή κύριε Τσόλος. Έχουμε εδώ μια αλλαγή πρακτικής που ξεκίνησε με τον Κίνοκαν, δεν απατώμε. Ε, πιστεύω ότι πρέπει πλέον ο Επίτροπος να λαμβάνει με την υπογραφή του την πολιτική ευθύνη για τις εκθέσεις αυτές. Το ίδιο ισχύει και με τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουμε, όπου έχουμε την αρμοδιότητα από την ε, νέα συνθήκη της Λισαβόνας και θέλουμε συγκεκριμένα να μας λέτε τα χρήματα τα οποία έχετε διαχειριστεί, πώς τα χρησιμοποιήσατε και με τι πολιτικό στόχο ε, αξιοποιήθηκαν. Τώρα έχετε συγκεκριμένους πολιτικούς ε, στόχους, πολλές φορές περίπλοκους, Στόχου οριζόντιου, ανάπτυξη υπαίθρου κτλ. Όχι τόσο στοχευμένους, το, όχι τόσο περιορισμένους και εστιασμένους όπως το παρελθόν. Θέλω λοιπόν να βλέπω στην εκθεσή σας εάν και πώς επιτύχατε τους στόχους που επιδιώκατε. Και επίσης κύριε Τσόλου θα ήθελα κάποιες ε, προτάσεις για αυτόματη διακοπή ή και πάυση των πληρωμών προς ένα κράτος μέλος το οποίο δεν ε, ε, συμμορφούνται προς υποχρεώσεις του. Μίλησα νωρίτερα για την Ελλάδα, δεν θα επαναλάβω το παράδειγμα αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε τι όνο. Επίσης θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερο για μηχανισμούς ελέγχου ή μάλλον διόρθωση. Μπορεί να έχετε καλού μηχανισμού διόρθωση και εποπτεία, αλλά πάλι κάποια ποσά συνολικά βλέπουμε ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως πρέπει. Θερυπίν. Από αυτά που μας λέει το 2006 το ελεγκτικό συνέδριο, 42% των ποσών ε, είναι αυτά που ανακτήθηκαν. Ε, καλά, καλά ποσοστά είναι για ανάκτηση των καταβλημένων. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι κακό ποσοστό, αλλά θα ήθελα να φτάσουμε στο 100% σε ανάκτηση. Επίσης για το 2009 έχουμε μόνο 10% ανάκτηση μόνο 10% ήταν τα ποσά τα οποία ανεκτήθησαν ενώ είχαν αχρεωστώς καταβληθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. 10% λοιπόν μόνο ποσά επεστράφησαν. Εσείς επίσης μιλάτε για τον περίφημο κανόνα 50-50, μισό-μισό. Αυτό σημαίνει ότι το 50% του ποσού που αχρεωστώς κατεβλήθη το καταβάλει το κράτος μέλος ως ποινή. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Αλλά, ένα λεπτό, εάν ακολουθήσουμε την λογική αυτή και δούμε ότι 10% επεστράφει μόνο και επίσης κατέβαλε το κράτος μέλος 50% ως κύρωση, τότε έχουμε χάσει 60% του συνολικού ποσού και το κράτος μέλος έχει επιπλέον καταβάλει ως ποινή, την οποία θεωρείται αιτιολογημένη πολύ καλά, ε, το 50%. Δηλαδή ο φορολογούμενος έχει έχει χρεωθεί δύο φορές. Αυτό δεν είναι λογική που να ικανοποιεί τη δική μου ε, τι σκοπιμότητε τι οποίε εγώ βλέπω σε αυτό το σύστημα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να διακόπτονται οι πληρωμές. Εφόσον κάποιος δεν ε, αποδεικνύει ότι έχει ορθά εισπράξει τα χρήματα, πρέπει να διακόπτεται η πληρωμή. Δεν έχει νόημα να επιβάλλονται τιμέ. Και στη συνέχεια βέβαια η πάυση. Επίση, ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η απλούστευση. Είπα και νωρίτερα ότι θα ήταν καλό να έχουμε μια κοινή ερμηνεία των κανόνων, ίσω όχι ε, μόνο το, ε, ε, δεν αρκεί όμως να έχουμε μόνο κανόνε, είναι απαραίτητο να είναι και σαφείς οι κανόνε και κατανοητοί οι κανόνε. Και έτσι θα ήταν καλό να ερευνήσουμε ποιοι είναι οι όροι για την εκτέλεση που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη, που έχουν εισαχθεί στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να δούμε πού χρειάζεται η απλούστευση, για να είναι σε 27 κράτη-μέλη οι ορισμοί μεν όπως είπαμε αναλογική, δηλαδή να λέμε ότι πράσινη έκταση είναι άλλο πράγμα στη Σκωτία, άλλο πράγμα στην ε, Βουλγαρία, αλλά από την άλλη να μπορούμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία της απλούστευσης σε όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν προτιμούν να προχωρήσουν στην απλούστευση γιατί μπορούν να ε, ε, υποκρύπτονται κάτω από τους περίπλοκους κανόνες και τη γραφειοκρατία. Ε, ότι αυτό ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να έχουμε προγράμματα δράσης απλά, προγράμματα δράσης τα οποία περιμένω και από εσά να δω το ταχύτερο και δει μέχρι την Άνοιξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι θέλετε, πρώτα η Κομισιόν και μετά το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, η Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, κύριε Χατζημαρκάκη για την παρουσίαση που κάνατε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αποσαφηνίσω κάποια στοιχεία και να σας δώσω και κάποια στοιχεία νέα. Όσον αφορά το Ajax, αυτό το ΩΣΔΕ, είναι ένα σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από την Κομισιόν τα τελευταία χρόνια και μπορώ να διαπιστώνω ότι και τον ένα χρόνο που είμαι στη θέση που βρίσκομαι τώρα, αλλά και γενικότερα διαπιστώνω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να ε, στηρίξουμε την, ε, ε, την γεωργική παραγωγή και notamment le contrôle des αρκεί να διατηρήσουμε την, ε, την μη σύζευξη των ε, πολιτικών και των ε, δαπανών. Πρόκειται για ένα σύστημα, αυτό το ΩΣΔΕ είναι ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα αγροτεμάχια και τα δεδομένα με τους γεωργούς. Το 2009 καταφέραμε να καλύψουμε παραπάνω από το 80% των ε, γεωργικών δαπανών ε, μέσω του ΟΣΔΕ και καλύπτεται έτσι και ένα μέρος του προγράμματος και του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή της ανάπτυξης της ε, υπαίθρου και εκεί περιλαμβάνονται και περιβαλλοντικές δράσεις. Επομένως καλύπτουμε ολοκληρωμένα τον πρώτο πυλώνα και εν μέρη και τον δεύτερο ε, πυλώνα. Μπορούμε επομένως στον πρώτο πυλώνα να έχουμε καλύτερα στοχευμένες δαπάνες και ελπίζουμε ότι στο μέλλον ο ΟΣΔΕ θα μπορέσει να αποτελέσει και μία ε, καλή βάση και για τον, για δεύτερο πυλώνα. Επίσης, είναι μια βάση η οποία μπορεί να βελτιωθεί, γιατί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχουμε στους ελέγχους στα κράτη-μέλη, αποφασίσαμε ε, να ε, οθήσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά την διαχείριση. Και το και το κέντρο ερευνών της ε, ε, Κομισιόν ε, δίνει κάποιες λύσεις κυρίως όσον αφορά την μέτρηση των αγροτομαχίων και δεν περιμένουμε επομένως πλέον να διαπιστώνουμε μόνο σαν έλεγχη της Κομισιόν τα προβλήματα αλλά πιέζουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν μόνα τους τους ελέγχους και να επιφέρουν βελτιώσεις μόνα τους. Είναι γεγονός ότι κυρίως όσον αφορά τα αγροτεμάχια έχουμε διαπιστώσει ελλείψεις και προβλήματα ε, όσον αφορά ε, τη βάση δεδομένων. Επίσης, ε, κάθε πέντε χρόνια λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα φωτογράφηση των αγροτεμαχίων ε, αλλά με τα κράτη-μέλη που έχουμε προβλήματα ζητούμε η επαναφωτογράφηση να γίνεται στα τρία χρόνια. Στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μπορεί συμπληρούμενο και βελτιούμενο να αποτελέσει έναν αντικειμενικό τρόπο ελέγχου του συστήματος ελέγχου επιτόπου των αγροτεμαχίων. Ε, μίλησατε για την ελληνική περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας όντως έχει άρει την επιφύλαξη ε, για την περίπτωση αυτή γιατί έχουμε μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά σαφής όσον αφορά ε, την ε, εμπλοκή των δαπανών, όσον αφορά τη δέσμευση λοιπόν των κονδυλίων. Στην ελληνική περίπτωση διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Ζητήσαμε λοιπόν πρόγραμμα δράσης το πρόγραμμα δράσης και υπό την απειλή της δέσμευσης και με την επιφύλαξη η οποία είχε μπει στην έκθεση πιέσαμε την ελλάδα έτσι ώστε να ξεκινήσει και να εφαρμόσει το σύστημα. από τη στιγμή λοιπόν που η χώρα ακολούθησε δεν είχαμε λόγο ε, να μην άρουμε την επιφύλαξη τώρα. Ε, το εάν θα λειτουργήσει μετά το σύστημα θα το δούμε αργότερα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε, ε, είναι διτή η προσέγγιση, από τη μία πλευρά έχουμε το εάν αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα και δεύτερον, εάν εφαρμοστεί σωστά. Εμείς ε, ε, ζητήσαμε την επιφύλαξη γιατί βρήκαμε ελλείψεις στο σύστημα. Από τη στιγμή που το σύστημα, η μεθοδολογία βελτιώθηκε όσον αφορά τον έλεγχο και τη φωτογράφηση των αγροτεμαχίων, δεν είχαμε λόγο να διατηρήσουμε την επιφύλαξη. Τώρα, ο ε, διοικητικός έλεγχος ο οποίος θα γίνει βάσει της βάσης δεδομένων εάν, εάν δείξει προβλήματα, εάν από αυτόν τον έλεγχο προκύψουν προβλήματα τότε θα δούμε ε, τι θα κάνουμε. Χαιρετίζω επίσης την πρότασή σας ε, ε, για το να δούμε το ενδεχόμενο όπως κάνουμε ε, και με την, ε, τις πολιτικές συνοχής το ενδεχόμενο λέω τριμερών συζητήσεων. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρως αναλαμβάνει τις ε, ε, υποχρεώσεις της αλλά είναι γεγονός ότι ε, πρέπει να μιλάμε και με τα κράτη-μέλη να δούμε πώς έχουν οργανώσει τους ελέγχους τους και ενδεχομένως θα ήταν μια καλή ιδέα να είναι παρόν και το ελεκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των, του ορισμού των γεωργών. Το είπα ήδη και στην αρχική μου παρέμβαση πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αποσαφινιστεί στο μέλλον. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κανονισμός του Συμβουλίου για τις άμεσες πληρωμές προβλέπει ότι γεωργός είναι αυτός ο οποίος εργάζεται στην υγεία ή, ε, ή όχι και ή τις διατηρεί σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Δεν λέει και λέει «ή». Είναι διαζευκτική η διατύπωση. Σύμφωνα λοιπόν με, τις, με τα λεγόμενα, με τα αναφερόμενα στον κανονισμό, τη στιγμή που έχουμε γεωργό ο οποίος καλλιεργεί τη γη ή γεωργό ο οποίος διατηρεί τα αγροτεμάχια του σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση τον θεωρούμε γεωργό. Το, ο σκοπός είναι και για το μέλλον βέβαια να διατηρήσουμε μονάχα υπό τον όρο γεωργός αυτούς που πραγματικά ενεργητικά ασχολούνται με την γεωργία. Ε, τώρα υπάρχει και η περίπτωση ε, των γεωργών οι οποίοι είναι ε, οι αγρότες του καναπέ, οι sofa farmers. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αφηνήσουμε. Να σας πω επίσης ότι έχουμε διαδικασίες αρκετά ε, σαφείς όσον αφορά την δέσμευση των ε, κονδυλίων. Το μπλοκάρισμα λοιπόν των ε, πληρωμών το χρησιμοποιούμε εμείς κυρίως σαν προτροπή προς τις χώρες έτσι ώστε να συμμορφωθούν. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να κρατήσουμε τα χρήματα, εμείς θέλουμε να πιέσουμε τις χώρες να βελτιώσουν το σύστημα, να προχωρήσουν διαρκώς βελτιούμενες. Ε, μέχρι τώρα αυτή η απειλή την οποία κραδένουμε, ε, την οποία χρησιμοποιήσαμε για τη Βουλγαρία και την ε, Ρουμανία, λειτουργήσε για την ώρα καλά. Το χρησιμοποιήσαμε στην Ελλάδα, δεν χρειάστηκε όμως τελικά να παίξουμε το χαρτί αυτό, γιατί η Ελλάδα προσαρμόστηκε, συμμορφώθηκε. Ε, τώρα, για τις δύο περιπτώσεις που ανέφερα προηγουμένως, έχουμε ένα σχέδιο δράσης. Και εγώ βεβαίως θα θέσω σε εφαρμογή την απειλή τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, εάν δεν συμμορφωθούν οι χώρες. Ε, στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και στον νέο χρηματοδοτικό κανονισμό θα δούμε τι θα κάνουμε με τις πληρωμές. Αλλά πάντως πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προτρεπτικό τρόπο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σας ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να υπογράφουν μία εθνική δήλωση έτσι ώστε να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ε, ευθύνη. Αλλά πέρα από την ε, υπογραφή του Υπουργού θα πρέπει να γίνεται και ένας έλεγχος. Η ιδέα να ζητούμε από τον οργανισμό πιστοποίησης ή έναν άλλον ανεξάρτητο οργανισμό να ελέγχει τον οργανισμό που κάνει τις πληρωμές μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια σαφέστερη άποψη για το τι ισχύει επιτόπου. τόπου. Τελευταίο σημείο όσον αφορά την ανάληψη ευθύνης των επιτρόπων. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην αναλάβω τις ευθύνες μου. Ξέρετε όμως ότι από τη σύστασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της σαν κολέγιο και επομένως δεν μπορώ εγώ εξ ονόματος της Επιτροπής αλλά με το δικό μου όνομα να υπογράψω κάποια δήλωση ε, θα πρέπει να, ε, ολόκληρο το κολέγιο των επιτρόπων να αποφασίσει ή να υπογράψει ε, και επομένως αυτό συμβαίνει και με την παρούσα έκθεση. Όσον αφορά τώρα τις επιστροφές, τις ανακτήσεις κονδυλίων από τη στιγμή της εφαρμογής ε, του κανόνα 50-50 και που δεν την έχουμε, τον έχουμε εφαρμόσει τον κανόνα αυτό για να πληρώσει ακόμα περισσότερα ο φορολογούμενος. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν από τις εφαρμογής αυτού του κανόνα 50-50. Οι ανακτήσεις από πλευράς κρατών μελών έχουν αυξηθεί. Για το 2007 είχαμε 33% ανάκτηση ε, και εφαρμόζουμε λοιπόν ε, από την τέταρτη χρονιά τον κανόνα του 50-50. Αλλά όπως υπάρχει αυτή η απειλή του 50-50, για το 2007 είχαμε εξέλιξη. Από το 33% φτάσαμε στο 49% για το 2009 ε, και παραμένει βεβαίως το 51% για το οποίο εφαρμόζουμε τον κανόνα 50-50 και αν συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε ο κανόνας 50-50 βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών για ενίσχυση του συστήματος ανάκτησης είναι πολύ μεγαλύτερο. Για το 2008 από το 24% περάσαμε στο 40% τη δεύτερη χρονιά. Επομένως μπορούμε να αναμένουμε ότι τον τρίτο χρόνο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάκτηση. Και επίσης για το 2009 έχουμε 24% ε, ποσοστό ανάκτησης. Πιστεύω ότι και εδώ μπορούμε και πρέπει να έχουμε ε, βελτιώσεις, ε, να πλησιάσουμε και στο 100%. Πάντως πιστεύω ότι και εδώ εμπλέκεται και η ευθύνη των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί διάφορα προτρεπτικά μέτρα. Ε, σε... Όσον αφορά την απλούστευση το έχω πει και το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Αποφάσισα να δημιουργήσω αυτή την ad επιτροπή με ε, εμπειρογνώμονες οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα, γνωρίζουν την κατάσταση επιτόπου και οι οποίοι θα δουλέψουν την μεταρρύθμιση μαζί με την ε, νομοθετική δέσμη έτσι ώστε ε, το αποτέλεσμα των μελετών να μην έχει αρνητική επίπτωση επιτόπου και στους ενδιαφέραμους. Ευχαριστώ πολύ. Το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω τρία σημεία. Καταρχάς την απλούστευση κατά δεύτερο λόγο τις τριμερείς πληρωμές και κατά τρίτο λόγο τις ανακτήσεις. Ως προς την απλούστευση. Προφανώς το ελεκτικό συνέδριο συμφωνεί. Θα πρέπει οι κανόνες να είναι πιο απλοί, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη κατά την εφαρμογή, την υλοποίηση των συγκεκριμένων ε, δράσεων και λειτουργιών. Αν είναι πιο απλοί οι κανόνες, τότε ε, λάθη θα προκύπτουν από, από λιγότερο αριθμό πηγών. Πολύ συχνά περιπλέκονται τα πράγματα γιατί τα κράτη-μέλη υποβάλλουν περαιτέρω επιπρόσθετα αιτήματα και ή μάλλον θα έλεγα περιπλέκονται τα πράγματα γιατί πέρα από τις ευρωπαϊκές διατάξεις υπάρχει και η εσωτερική νομοθεσία εσωτερικές διατάξεις των κρατών μελών και έτσι η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη. Έχουμε την έκθεση για τους όρους που θα πρέπει να πληρούνται. Έκθεση δική μας του ελεγκτικού συνεδρίου. Και εκεί κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την πολιτική της πολλαπλής συμμόρφωσης. Επίσης, εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συστάσεις, κάτι το οποίο είπε και ο κ. Επίτροπος για να απλουστευτεί ο ορισμός, η έννοια του δικαιούχου και η έννοια της ε, γεωργικής δραστηριότητας, ώστε να ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος της ενίσχυσης. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι το παράδειγμα που ανέφερα, για παράδειγμα ε, μια έκταση 530 εκταρίων, που ανέφερα στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Αυτό ήταν σφάλμα και παραμένει σφάλμα. Ορισμένα μέρη αυτής της, έκθεση, ε, της έκτασης είχαν διατηρηθεί σε καλή γεωργική κατάσταση, δεν ήταν όμως επαρκής ο αριθμός τους, δεν ήταν αρκετά. Επομένως, το σύνολό τους αυτά τα αγροτεμάχια είχαν ε, λάβει εσφαλμένα αν θέλετε ε, την δυνατότητα το δικαίωμα για ενιαία άμεση ενίσχυση δεν ήταν όλα, όλες οι εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση, το σύνολο. Ε, και αυτό το αναγνώρισαν οι επίσημες αρχές ε, της Βουλγαρίας. Δηλαδή η ίδια η κρατική αρχή αναγνώρισε την ύπαρξη σφάλματος στην περίπτωση αυτή, στο παράδειγμα αυτό. Η απλούστευση δηλαδή θα μας ε, κάνει να αποφύγουμε τα σφάλματα, αλλά όχι όλα. Αυτά για την απλούστευση. Τώρα, ως προς το θέμα ε, των τριών μερών. Κυβέρνηση, Κομισιόν και Ελεκτικό Συνέδριο. Το Ελεκτικό Συνέδριο στέλνει τις παρατηρήσεις στο κράτος μέλος πάντοτε και κοινοποιεί τις παρατηρήσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως είναι ενήμερη και το κράτος μέλος και η Επιτροπή. Το ελεγκτικό συνέδριο πηγαίνει επί τόπου, στέλνει τις παρατηρήσεις στο κράτος μέλος και στέλνει και αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κάθε μετά απαντά. Υπάρχει δηλαδή αυτή η τριμερής διαδικασία. Αυτό το οποίο δεν γίνεται είναι εκπρόσωποι να συσκεφθούν στο ίδιο δωμάτιο, στην ίδια αίθουσα. Αλλά και να γίνει τέτοιου είδου σύσκεψη δεν θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία γιατί το σημαντικό είναι να πηγαίνει κανείς επί τόπου ε, για να εντοπίζει το πρόβλημα και να βρίσκει και λύσεις. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι παρατηρήσεις μας είναι σωστά τεκμηριωμένες και δεν το αναγνώρισε επειδή ε, συσκεφθήκαμε μαζί μέσα σε μια αίθουσα, αλλά επειδή μετέβη επιτόπου και διαπίστωσε του λόγου του αληθές. Θα ήθελα λοιπόν να το επαναλάβω αυτό, ότι αυτή η τριμερής εξέταση της κατάστασης ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επομένως, η βασική μας, η αρχική μας έκθεση ε, καταρτίζεται μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπάρχει αυτή η αντίφαση αν θέλετε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τις απόψεις των κρατών μελών, ωστόσο ο τελικός διάλογος, η τελική συζήτηση αν θέλετε για το κατά πόσο είναι τεκμεριωμένες οι παρατηρήσεις γίνεται μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο τελικός υπεύθυνο αν θέλετε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τέλος, ως προς τις ανακτήσεις ε, θα έλεγα ότι θα ε, δημοσιεύσουμε μια έκθεση λεπτομερή για το θέμα των ανακτήσεων όπου θα γίνεται πλήρη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και θα περιβάλλονται και συστάσεις για τη βελτίωση. Ε, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες γιατί ε, θα γίνουν πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Ευχαριστώ συνάδελφος κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πετροβά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Όπως είπατε στην αρχή, η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη μία από τις πολιτικές που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών. Και γι' αυτό μας απασχολεί πολύ συχνά εδώ στην Κοκομπού. Το ποσοστό σφάλματος είναι λίγο υψηλότερο από το 2%. Άρα δεν έχει περάσει ακόμη στην πράσινη ζώνη γεωργική πολιτική. Μάλιστα, ο εισηγητή μας ανέφερε ότι στην ετήσια έκθεση της ε, Γενικής διεύθυνση για τη Γεωργία 735 εκατομμύρια ευρώ δεν διατίθενται, 42 δηλαδή τα ποσά που χρειάζεται να ανακτηθούν Βέβαια αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2006 που είχαμε αντίστοιχα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς ανάκτηση. Τα ποσοστά λοιπόν είναι αρκετά καλά στην ανάκτηση 50% σε άλλα κράτη χαμηλότερο Ερωτώ λοιπόν πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει, να πείσει τα κράτη, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή. Επίσης, η απλούστευση των διαδικασιών. Τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασιών. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ε, γίνει εις βάρος της ποιότητας των ελέγχων. Πώς λοιπόν μπορεί να εξασφαλιστεί η λεπτή αυτή ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της ποιότητας. Απλούστευση διαδικασιών, ποιότητα ελέγχων. Ο κύριος Τσόλος. Όσον αφορά την ανάκτηση, βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όπως είπα νωρίτερα όμως, διαπιστώνουμε ότι με τον κανόνα 50-50 τώρα τα κράτη-μέλη έχουν κίνητρο να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάκτησης. Ιδάλλως επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός τους ευθέως. Και γι' αυτό με τον κανόνα αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολύ πιο στενά τα κράτη-μέλη και όταν επιστώνουμε προβλήματα ε, τα πιέζουμε περισσότερο. Δεν θέλω όμως να μιλήσω μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, γιατί είναι μοιρασμένη η ευθύνη. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δική, το δικό του μερίδιο ευθύνη, το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι και στον, τον εθνικό φορολογούμενο για το πώς διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό τους. Στον κανόνα 50-50 λοιπόν βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη όντως έχουν πολύ περισσότερα κίνητρα να ε, επιταχύνουν τη διαδικασία ανάκτησης. Για την απλούστευση. Συμφωνώ. Άλλωστε, το διαπιστώνω και εγώ όταν ε, πηγαίνω στην ε, Κομάγκρη μου λένε πάντα ότι χρειάζεται απλούστευση το δυνατόν προς των κανόνων. Αυτό που τους λέω εγώ είναι ότι, σαν απάντηση είναι ότι δεν μπορεί αυτή η απλούστευση να αποδυναμώσει τα συστήματα των ελέγχων. Και έτσι λοιπόν, παραλίλου με την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου, με το ΟΣΔΕ, αλλά και με ένα προσωπικό υψηλής κατάρτισης που θα υλοποιεί τους ελέγχους αυτούς. Θέλω στην ε, μεταρρύθμιση τώρα της γεωργικής πολιτικής να ακολουθήσω ακριβώς αυτές τις δύο, τους δύο διάβλους, δηλαδή την ε, υποχρέωση για τον γεωργό ε, να πληρεί τι προδιαγραφέ και του σεβασμού του περιβάλλοντο και τη ευημερία των ζώων κτλ. Αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι βάσει των οποίων μπορεί να υλοποιήσει αυτέ τι προδιαγραφέ. Γι' αυτό θέλω με βάση την νομοθεσία να προχωρήσω προ πρακτικού οδηγού που μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει, να ενημερωθεί ο γεωργός, ο ίδιος, αλλά και η υπηρεσία που θα του προσφέρει τις συμβουλές και ο ελεγκτής επίσης ο οποίος θα κληθεί να τον υλοποιήσει. Να γνωρίζει δηλαδή και ο ελεγκτής τι πρέπει να ελέγξει και πώς θα διαπιστώσει ότι τηρήθηκε ο κανόνας. Και επίσης θέλουμε μια καλύτερη χρήση τη άμεση ενίσχυση, να τη συνδέσουμε, να συνδέσουμε αυτές τις ενισχύσεις με στόχους σαφείς και να προσδιορίσουμε ποιο θα είναι ο δικαιούχο, ποιο θα είναι ο τύπο του δικαιούχου καλύτερα και υπό ποιου όρου θα διατίθεται η ενίσχυση. Και αυτό όπως συζητήσαμε μόλις τώρα, ακόμη και αν ε, σε περίπτωση όπως αυτή της Βουλγαρίας έχουμε από την φωτογραφική ε, παρακολούθηση μία καλή εικόνα ενός ε, αγροτεμαχίου. Έχουμε ένα αγροτεμάχιο το οποίο έχει παρουσιάσει μια καλή εικόνα ήταν επιλέξιμο για ε, χορτολιβαδική έκταση καλύτερα, ήταν επιλέξιμο για ε, ενίσχυση, παρότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ίχνη περάσματο ζώων κτλ. Και, και χωρίς να έχει εμπλακεί ο ίδιος ο ε, σε βλέπουμε ότι είχε καλή εικόνα, ικανοποιητική εικόνα αυτή η χορτολιβαδική έκταση. Ευχαριστώ πολύ. Βον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω ε, φαίνεται ξεκάθαρα στην έκθεση είναι ότι καταγράφονται υπερβολικά πολλά επιλέξιμα τεμάχια, αγροτεμάχια, χορτολιβαδικές εκτάσεις. Γι' αυτό νομίζω έχουμε πρόβλημα στους ορισμούς. Πρέπει να προσδορίσουμε τι σημαίνει επιλέξιμη γη, πρέπει να, σημαίνει, να ορίσουμε τι σημαίνει ε, δραστήριος ε, γεωργός είχατε πει στην ετήσια σας έκθεση ότι θα δώσετε τέτοιους ορισμούς. Πούντι. Θα πρέπει να περιμένουμε για την επόμενη μεταρρύθμιση μετά το 2013 της ε, κοινής πολιτικής. Τα συστήματα εποπτείας. Ναι, όντως, όπως το είναι και σημαντικά, αλλά ε, εμείς φερειπίν στην Ουαλία τώρα θα περάσουμε σε ένα ψηφιακό σύστημα θα είναι πολύ πιο ακριβής η μέτρηση και ο υπολογισμός των εκτάσεων. Έχετε εσείς αντίστοιχα πρόθεση ε, να ε, επεκτείνετε τα ψηφιακά μηχανογραφημένα συστήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζω αυτό θα βοηθήσει πολύ. Απάντηση, Τσόλος για τους ορισμούς ε, ποιο, του ποιος ε, γεωργός είναι δραστήριος και ποια γη είναι επιλέξιμη. Αυτό στηρίζεται σε κανονισμό του Συμβουλίου. Τώρα θα έπρεπε να ήταν κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου με τη νέα ε, συνθήκη. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία μεταρρύθμισης κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί μετά το 2013. Ακόμη και τώρα λοιπόν να κάναμε τροποποίηση του κανονισμού ή να ξεκινούσε μάλλον τη διαδικασία ε, για τροποποίηση του κανονισμού είναι τέτοιε οι διαδικασίε σε επίπεδο Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που δεν θα ήταν πιο σαφείς οι ε, ορισμοί, δεν θα είχαμε μάλλον του οδηγούς πριν το 2013. Άρα χρόνο δεν θα κερδίσαμε, μόνο θα είχαμε δύο παράλληλες διαδικασίες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμο. Θεωρούμε ότι είναι πιο σκόπιμο να ενταχθεί αυτή η νέα ιδέα με τους ορισμούς κτλ. στη συνολική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έτσι ώστε να έχουμε ε, να την εισαγάγουμε μαζί με, την, ε, με τις άμεσες ενισχύσεις. Με το νέο σύστημα μάλλον. Επίσης, βάση των δεδομένων ε, για αυτά τα αγροτεμάχια και χαρτολιβαδικές εκτάσεις είναι όντως ψηφιοποιημένες γιατί γίνεται η φωτογράφηση από το δορυφόρο και η οριοθέτηση των ε, τεμαχίων ε, των κλήρων γίνεται ψηφιακά. Εσεί όμω αναφέρεστε σε κάτι άλλο, σε ένα ψηφιακό σύστημα ταυτοποίηση ζώων που έχει εισαχθεί στην ε, ε, Ουαλία. Όπω έχουμε παραδείγματι και για τι προβατίνε ήδη. Το ΩΣΔΕ συνδέεται με ένα σύστημα πέραν αυτό των εκτάσεων και των γεωργών, με ένα σύστημα λοιπόν ψηφιακό ζώων, καταχώρηση ζώων. Και υπάρχει δυνατότητα ε, ανάγνωσης ψηφιακής αυτού του μητρώου ε, των ζώων. Θα μπορούσε και αυτό να εισαχθεί. Αλλά πάντως ε, η ψηφιοποίηση των εκτάσεων έχει ήδη γίνει. Βεβαίως υπάρχουν κράτη τα οποία κάνουν ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταγραφή των μεγάλων εκτάσεων, των μεγαλύτερων, με τι οποίε μπορεί να υπάρχουν περισσότερε εκμεταλλεύσει. Κάποια άλλοι έχουν περάσει στην ε, καταγραφή τη συγκεκριμένη εκμετάλλευσης που χρησιμοποιεί ένα γεωργό. πιο συγκεκριμένα δηλαδή. Αλλά πάντως το ψηφιακό σύστημα υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Μιούλντερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, κυρίως ε, αυτή που αφορά την απλούστευση των κανόνων και των κανονισμών. Αρκετά χρόνια πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε ε, μία έκθεση για την απλούστευση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ε, ε, έτσι ώστε αν κάποιος ας πούμε παράγει γάλα πριν στο ιδιωτικό τομέα αναφέρομαι τώρα εάν ε, μια βιομηχανία θα αγοράσει το γάλα θα κάνει επιπλέον ελέγχους. Επομένως το κράτος μπορεί να κάνει ε, τους ελέγχους αλλά μερικές φορές ε, γίνεται ο έλεγχος δύο φορές. Δηλαδή η ιδιωτική επιχείρηση, το ιδιωτικό εργοστάσιο κάνει κάποιους ελέγχους και μετά το κράτος κάνει αντίστοιχους ίδιους ελέγχους. Λέγαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο οι έλεγχοι έτσι ώστε να μην ε, γίνουν ε, οι τόσο ε, ανώφελοι διπλή έλεγχοι. Κάτι άλλο τώρα. Διπλός, διπλή νομοθεσία. Εάν έχετε σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφούστε προς, τη, προς τους κανονισμούς και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. αλλά το ποσοστό εφαρμογής καμιά φορά δεν είναι ικανοποιητικό γιατί υπάρχουν και αντιφάσεις. Ας πούμε, η οδηγία για τα, φωσφορούχα ε, του 90, η οποία αντιτίθεται από την αντίστοιχη οδηγία του 2007. Ας πούμε, στην πρώτη οδηγία αναφέρεται ότι πουθενά στην Ευρώπη με πολύ ελάχιστες εξελίξεις δεν μπορεί κανείς να έχει ε, πάνω από ένα ml ε, ε, ε, ανά εκτάριο ενώ σε άλλες, στην άλλη περίπτωση αναφέρεται ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχει κανείς παραπάνω από 50 ml μιλιγκράμμ φωσφάτων. Και αυτό βεβαίως κάνει πολύ περισσότερα ε, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανά εκτάριο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί στην πρώτη οδηγία αναφέρεται ότι δεν μπορεί να έχει κανείς παρουσία φωσφάτων ε, πάνω από 1,7. Ε, εδώ έχουμε αντιφατική νομοθεσία. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, όσον αφορά, απάντηση του Επιτρόπου, όσον αφορά την ε, απλούστευση, ναι, ε, όντως θα μπορούσε να υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις μονάχα εν μια μορφή πιστοποίησης. Από τη μία πλευρά όμως ελέγχουμε την, ε, το, την ποιότητα του ε, γάλου, αλλά, του γάλακτος, συγγνώμη. Αλλά αυτό δεν είναι αντικειμενικός έλεγχος όσον αφορά τις δικές μας απαιτήσει. Ε, σχετίζεται με την ε, τιμή του γάλακτος. Και ούτως ή άλλως αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται για κάποιο δημόσιο οργανισμό. Αυτό αυτός ο έλεγχος γίνεται από την ίδια τη γαλακτοκομική μονάδα έτσι ώστε να επιτύχει καλύτερη τιμή. Ε, σχετίζεται με την ε, ιδιωτική αγορά και επομένως είναι δύσκολο ε, να συνδέσουμε την ποιότητα με έναν δημόσιο έλεγχο. Όσον αφορά τώρα την πολλαπλή συμμόρφωση μιλάμε για την εφαρμογή όντως ενός ευρωπαϊκού κανονισμού. Όσον αφορά τώρα για την, για την άλλη σας ερώτηση, η απλούστευση προς την οποία εμείς ε, εργαζόμαστε και συνεργάζομαι και με τους συναδέλφους Ποτόσκι και Νταλή, δηλαδή για τους συναδέλφους του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, είναι να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε, να μεταφράσουμε τις ε, οδηγίες αυτές οι οποίες είναι πολύ τεχνικές για την ώρα να τις μεταφράσουμε λέω σε συγκεκριμένες δράσεις ε, που θα μπορούν να πιστοποιήσουν και να μετρήσουν μέχρι έναν βαθμό οι ίδιοι οι γεωργοί. Βεβαίως λέμε ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η νομοθεσία, αλλά η μέθοδη εφαρμογής της νομοθεσίας να γίνει πιο σαφής και πιο απλή ε, επιτόπου. Όσον αφορά τώρα τα φωσφάτα, εγώ δεν είμαι κοιτάξτε, εγώ δεν ε, ξέρω τι ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, αλλά ε, η χρήση των ε, αζωτούχων μπορεί να γίνει στην επιφάνεια, αλλά μπορεί να γίνει και πιο στο βάθος. Ο κίνδυνος όμως για την γεωργία σχετίζεται με τη μόλυνση των υδάτων επιφανείας Γι' αυτό ακριβώς ε, αναφερόμαστε περισσότερο σε τι είδους εντομοκτώνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ζανιοκτώνα κτλ. Οι εμπειρογνώμονες του περιβάλλοντος ασχολούνται με αυτά και αποφασίζουν τα ποσοστά και τις τιμές. Εγώ σαν Επίτροπος Γεωργίας πρέπει να διασφαλίσω ότι οποιοδήποτε είναι οι κανονισμοί τους εφαρμόζουν ε, οι γεωργοί έτσι ώστε να ξέρουν και καλύτερα και εδώ μπορώ να απλουστεύσω τα πράγματα, να ξέρουν οι γεωργοί τι πρέπει να κάνουν. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτησης. Έχουμε έναν πολύ καλό επίτροπο εδώ στην αίθουσα, έναν εξαιρετικό ε, ε ένα εξαιρετικό στέλεχος του ελεκτικού συνεδρίου, αναφέρομαι στον κύριο Κρέτεα, ε, ασχολείστε πολύ εντατικά με αυτό το φάκελο και σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Έχω κάποια ερωτήματα ωστόσο να απευθύνω και στον κύριο Κρετά και στον κύριο Επίτροπο. Ε, πρώτα στον κύριο Κρετά. Ως προς τη δειγματοληψία, το, το δείγμα το 2007 ε, είχατε περίπου 47, ε, 240, το 2007 είχατε ελέγξει κάποιες ε, ε, λειτουργίες και ο αριθμός αυξήθηκε τα επόμενα χρονιά. Την επόμενη χρονιά έχουμε λοιπόν 241 ελέγχους και επίπεδο αξιοπιστίας 95%. Αυτά τα νούμερα ε, συμμορφούνται με, τους, ε, με τα διεθνή πρότυπα. Νομίζω ότι είναι λίγα ως δείγματα. Είναι μικρός ο αριθμός των δειγμάτων, όποιος και αν ήταν αυτός αναέτος και γενικώ η γεωργία ήταν το ίμιση των δαπανών για το 2009. Σε γενικές γραμμέ, αυτή είναι μια γενική διαπίστωση. Τα συμπεράσματά σας, τα απορίσματά σας για το γεωργικό τομέα, για το επίπεδο ουσιώδων λαθών και σφαλμάτων, πώς συνδέονται τελικά με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που λέει ότι χωρίς επιφύλαξη πιστοποιούμε και αποδεχόμαστε τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύψετε τις ε, ε, ανταλλαγές απόψεων που είχατε στο εσωτερικό του οργάνου σας, αλλά πώς εξηγείτε από τη μία χωρίς επιφύλαξη να δέχεστε ε, τους τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη να υπάρχουν ουσιώδη λάθη ε, στο Γεωργία που είναι το 5% του προπολογισμού. Στρέφουμε τώρα προς τον κύριο Επίτροπο και θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή: ε, μιλούμε για την κοινή γεωργική πολιτική και ε, είναι ουσιώδης Όντως. Ε, μιλούμε επίσης για τις εθνικές δηλώσεις. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι αξιόπιστες. Έχω προτείνει ε, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να μας διαβεβαιώσουν ε, για το επίπεδο των ανεξάρτητων ελέγχων. Δεν θα πίστευα προσωπικώς αυτά τα οποία δηλώνουν τα κράτη-μέλη, η, κεντρική αρχή αν θέλετε. Επομένως, μπορείτε εσείς κύριε Επίτροπε να πιστοποιήσετε ότι αυτά τα όργανα πιστοποίησης είναι όντως ανεξάρτητα. Ότι είναι ανεξάρτητες οι αρχές που ε, πιστοποιούν ε, ε, τα τεκτενόμενα. Εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι οργανισμοί πιστοποίησης να ενταχθούν, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή ιεραρχία. Δηλαδή, δικά μας τελέχη να μεταβούν ε, στους οργανισμούς αυτούς πιστοποίησης. Να αποσπαστούν εκεί έτσι ώστε να ε, ξεφύγουν αυτοί οι οργανισμοί από την ε, ιεραρχία την διοικητική των κρατών μελών και να βελτιωθεί έτσι η αξιοπιστία τους, να είναι πιο ανεξάρτητος ως αρχές. Ο κύριος Κρετά, να σας απαντήσω για το δείγμα και για τις δηλώσεις. Τώρα, ως προς το δείγμα, ναι, έχουμε, αποφασίζουμε ένα συγκεκριμένο δείγμα, με έναν αριθμό δεγμάτων. Εκατομμύρια πληρωμές γίνονται συνολικά. Η στατιστική θεωρία μας λέει η βασική αρχή δηλαδή που χρησιμοποιούνται και στις έρευνες που γίνονται, στις έρευνες αγοράς, στις έρευνες της κοινή γνώμης, ότι αν πάρουμε ένα μικρό δείγμα και τους ζητήσουμε την άποψή τους, τότε θα μάθουμε την άποψη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων στη συνέχεια. Δηλαδή με μικρό αριθμό συναλλαγών ή λειτουργιών που διαλέγονται, επιλέγονται τυχαίω, μπορούμε να έχουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα για μεγάλο αριθμό πληρωμών. Τι μπορούμε να πούμε δηλαδή σε γενικές γραμμές με δύο λόγια. Ο αριθμός των δειγμάτων φτάνει σε ένα κατόφλι, σε ένα πλαφόν αν θέλετε και όσες πληρωμές και αν έχουν γίνει συνολικά ε, θα έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δηλαδή, σύμφωνα με την θεωρία, με 300 δείγματα ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, να είμαστε αρκετά πεπισμένοι ε, ότι θα έχουμε αντιπροσωπευτική εικόνα είτε έχει γίνει συνολικά ένα εκατομμύριο πληρωμές είτε έχουν γίνει συνολικά πέντε εκατομμύρια. Με τα 300 δείγματα βάσει της θεωρίας έχουμε επαρκή αριθμό δειγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο να παίρνει 300 δείγματα. Για το σύνολο των τομέων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για όλους τους ε, τομείς αν θέλετε. Είπατε ότι η Γεωργία ε, αντιπροσωπεύει το 50, άρα όντως πρέπει να κάνουμε περίπου 180 στα 360 δείγματα. Δεν, δεν πήραμε 180 δείγματα, πήραμε παραπάνω, πήραμε 240 δείγματα για να αυξήσουμε την αξιοπιστία του δείγματος αυτού. Δηλαδή, το συμπέρασμα και η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι αυτό το νούμερο, τα 241 δείγματα, ε, αρκεί, επαρκεί για να έχουμε ε, μια σιγουριά της, της τάξης του 95% στα συμπεράσματά μας. Παρόλα αυτά, από την επόμενη χρονιά τα γεωργικά θα τα χωρίσουμε σε πρώτο πυλώνα και σε δεύτερο πυλώνα και θα έχουμε δείγματα για κάθε πυλώνα ξεχωριστά. Δηλαδή θα γίνουν δύο δειγματοληψίες Άρα ο αριθμός των συναλλαγών, αν θέλετε, που θα εξεταστεί θα αυξηθεί και έτσι θα έχουμε επιπρόσθετη εξασφάλιση και σιγουριά, αν θέλετε. Αλλά ήδη με τον αριθμό των δειγμάτων βάσει της στατιστικής θεωρίας μπορούμε να είμαστε βέβαιοι κατά 95% ε, για τα ευρήματά μας, για τα ευρήματα των ερευνών μας. Αυτό καταρχάς. Τώρα, ως προς τις εθνικές δηλώσεις και την αξιοπιστία τους να σας πω το εξής. Βάσει της συνθήκης, το ελεκτικό συνέδριο καλείται ε, να ε, ε, αποφανθεί για την αξιοπιστία με βάση δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, η συνθήκη ζητεί από το ελεκτικό συνέδριο να αποφανθεί καταρχάς για την αξιοπιστία των λογαριασμών, ότι δηλαδή τα νούμερα είναι τα σωστά νούμερα στους λογαριασμούς, True and fair, λέει η συνθήκη. Δηλαδή μια δίκαιη, ε, πιστή απεικόνηση. Ε, πιστή λοιπόν απεικόνηση των συναλλαγών και της κατάστασης, εμπασχευτώς των ευρωπαϊκών λογαριασμών στο τέλος της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Αυτό ε, είναι το νόημα της αξιοπιστίας. Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα η το αίτημα περιορίζεται σε αυτά. Βάσει της συνθήκης δεν μιλούμε όμως εμείς για αξιοπιστία μόνο, μιλούμε και για ε, την, ε, το νομότυπο. Το ότι οι συναλλαγές ε, πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Έγιναν διάφορες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε θέση να πούμε ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι λογαριασμοί που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιόπιστοι από τη λογιστική λογιστική σκοπιά, βάση λογιστικών προτύπων. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, οι συναλλαγές είναι νομότυπες. Και εκεί τι λέμε. Αυτό είναι το δεύτερο που καλούμαστε να πούμε. Είναι νομότυπες και λέμε όχι, δεν φαίνονται ε, προς το παρόν ως προς ε, το Ταμείο συνεχή και τα κονδύλια που δίδονται στη Γεωργία. Δηλαδή, όντω είναι πιστή απεικόνηση, από την άλλη έχουμε απόσταση να καλύψουμε ω προ το νομότυπο των λογαριασμών. Δηλαδή υπάρχουν δύο σκέλη και ελπίζω να σα ε, το διευκρίνησε επαρκώ το θέμα. Ο επίτροπο κύριο Τσιόλο να απαντήσει τώρα. Τώρα, ω προ του οργανισμού πιστοποίηση. Θα σας απαντήσω ε, με βάση την αρχή της μοιρασμένη διαχείρισης ε, των κονδυλίων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένες ευθύνες, αλλά και το κράτος μέλος, το εκάστοτε, έχει ευθύνες. Τελική ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όντω. Αλλά το κράτος μέλος καλείται να αναλάβει τις ευθύνε του. Εάν οι οργανισμοί πιστοποίησης ε, τεθούν υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι αποδυναμώνουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει το κράτος μέλος στη διάθεσή του για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν ως ε, κράτος μέλος. Μπορούμε να ενισχύσουμε τους οργανισμούς πιστοποίησης, παρόλο που ε, ε, θα συνεχίσουν να παραμένουν υπό την εθνική διοικητική αριαρχία και στο εσωτερικό του κράτους μέλους ο Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών ελέγχει ε, το Υπουργείο Γεωργίας. Και έχουμε και το ελεγκτικά συνέδρια που ελέγχουν ε, τις ε, κυβερνήσεις, την κεντρική διοίκηση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διευκρινίσουμε περισσότερο τα στοιχεία που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία αυτών των οργανισμών, ώστε οι οργανισμοί πιστοποίησης να μην έχουν ε, σχέσεις που δεν θα έπρεπε με τις αρχές που ε, διεκπαιρεώνουν τους πληρωμές. Όμως θα έλεγα ότι ο οργανισμός πιστοποίησης είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο στη διάθεση του κράτους μέλους και δεν θα πρέπει να το αποδυναμώσουμε το κράτος μέλος. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε βήματα για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία αυτού του οργανισμού. Η κυρία Γκρέσλε, παρακαλώ. Ασφαλώ. Χωρί τα μελη θα τα είχαμε πάει καλύτερα στην Ευρώπη, θα είχαμε προχωρήσει πολύ. Όμως έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα κρίσιμο που έχει να κάνει και με, τον, ε, με το ελεγχτικό συνέδριο, ποιον μπορούμε να εμπιστευτούμε. Για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι πολύ περιπλοκό. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο ακριβή στους λογαριασμούς τους, κάποια άλλη είναι λιγότερο Αυτά που είναι λιγότερο ακριβή τα βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας και πρέπει κάπως να τα πείσουμε. Κύριε Επίτροπε, θα σας έδωσα ακριβώς ασφαλώς κάποιο σημείωμα το προσωπικό σας, το προσωπικό που σας περιβάλλει, το τι θα κάνατε, τι θα απαντούσατε στην ερώτηση, τι θα κάνατε σε περίπτωση που ε, προχωρήσει η διαδικασία για την εκτέλεση κατά τρόπο ε, μη ικανοποιητικό για σας. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι θα θέλατε από πλευρά του Κοινοβουλίου. Εγώ δυστυχώ είμαι εισηγήτρια στο θέμα αυτό, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν βοήθεια από πλευρά σα. Θα ήθελα κάποιε ιδέε για το τι έχετε, τι έχετε επιτύχει στο τομέα τη γεωργία εσεί και το προσωπικό σα, συγκεκριμένα για την υλοποίηση των κανόνων και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τα οποία έχετε διαθέσει τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Γιατί χθε ακούσαμε κάποιες περιπτώσεις ε, με ε, ανεπιτυχή υλοποίηση, ανεπαρκή υλοποίηση και υψηλά ποσοστά ανάκτηση. Εμένα λοιπόν δεν με νοιάζει αν υπάρχει ποσοστό σφάλματος 1, 1,5 ή 2%. Με ενδιαφέρει να γίνεται σωστά η δουλειά και κυρίως στου τομείς όπου υπάρχουν εντοπίζονται οι δυσκολίες, Βουλγαρία, Ρουμανία, κράτη υποψήφια προς ένταξη, ιδιαίτερω θα ήθελα να δώσετε προσοχή. Και να ξέρετε ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον πολύ το θέμα αυτό. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν καλά, καλές επιδόσεις, υπάρχουν κράτη τα οποία δεν τα πάνε τόσο καλά και πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεβίνα. Ξέρουμε ότι είναι τελευταία διαδικασία για απαλλαγή που αναλαμβάνει στη σταδιοδρομία του, γιατί μετά θα φύγει με σύνταξη. Σα εύχομαι κάθε καλό και ευχαριστώ πολύ για την μέχρι τώρα συνεργασία. Στην επόμενη λοιπόν διαδικασία έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα σχετικό με επιδοτήσει, οι οποίε λόγω κάποιων δικαστικών αποφάσεων στη Γερμανία δεν μπορούν να καταβληθούν, δεν επιτρέπεται. Τι θα τι κάνετε αυτέ, λοιπόν, Πώ θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Και το ποσοστό 0,3, 0,2% ποσοστό σφάλματος που έχουν κράτη όπω η Γαλλία ή η Γερμανία. Να σα πω τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γίνεται μια άπελπης προσπάθεια να εξευρεθούν σφάλματα στη Γερμανία που να δικαιολογούν την ύπαρξη της ιερικής πολιτικής. Στη Βάδη Βουτεβέργη, παραδειγματί, υπάρχουν κάποιες περιοχές ε, που είναι πολύ μικρά τα αγροτεμάχια, διότι όπως προχωρούσε η κληρολομιά μιας οικογένειας, μοιράζονταν ε, τα αγροτεμάχια μεταξύ των πολλών παιδιών μιας οικογένειας, έτσι είναι όλο και πιο μικρές οι εκτάσεις. Και έτσι Ε, η εκμετάλλευση γίνεται συνεταιριστικά με τους γείτονες. Διαφορετικά δεν έχει καμιά αξία η καλλιέργεια της γης ή ε, η κτηνοτροφία. Αλλά βέβαια τα χρήματα θα τα εισπράξει εκείνος ο οποίος έχει επισήμως αναλάβει τη γεωργική δραστηριότητα, την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έστω και αν εναλλάσσονται ή συνεργάζονται στο με αυτό. Άρα εκεί υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος. Γιατί κάθε φορά θα πρέπει να γίνεται στην αίτηση ο κατακαιρματισμός του τεμαχίου, της, αγρο... αγροτικής εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να γίνει πάλι η μέτρηση κάθε χρονιά των ίδιων τεμαχίων που καταμετρήθηκαν και την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη χρονιά και θα καταμετρηθούν και την επόμενη. Έχουμε παρουσία επόπτη ή ελεγκτή στην περιοχή επί 39 ολόκληρε ημέρε για να βεβαιωθεί κάθε χρονιά ότι είναι σωστή, σωστός ο χωρισμό των τεμαχίων. Ρωτώ λοιπόν, δεν μπορούν με κάποιο τρόπο ε, να βρούνε μια λύση ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση τα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για την ίδια την περιοχή, το κρατήδιο, είτε για την κεντρική κυβέρνηση στο Βερολίνο, αλλά και η Κομισιόν επίση δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτή την κατάσταση. Τέτοιε λοιπόν περιπτώσει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τι αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει λύσει. Τρίτη παρατήρηση. Η νέα περίοδο τη κοινή πολιτική θα πρέπει ασφαλώς να δώσει περισσότερη έμφαση στην δυνατότητα ελέγχου τη στήριξη των διατάξεων. Αυτά τα οποία προβλέπετε να καταθέσετε ως προτάσεις λοιπόν για την νέα αυτή ε, περίοδο, για την νέα αυτή αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής, θα έχουν ιδέες για πιο αυστηρούς ελέγχους, για πιο αποτελεσματική εφαρμογή. Ο κύριος Επίτροπος, σχετικά σχετικά με την εκαθάριση των λογαριασμών Υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία τα οποία δεν συμμερίζεται με το συνέδριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερή έστω και αναδύναμη μείωση του ποσοστού λάθους όπως είπα και προηγουμένως, αυτό ε, οφείλεται και σε πρώτους ελέγχους που κάνουν τα ίδια τα κρατη επιτόπου, που ακολουθούνται από τους ε, ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το ποσοστό ε, το οποίο βαρύνει, το δαπανών που βαρύνει τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό ε, είναι σαφής και μετά από μελλοντική συμμόρφωση καθώς επίσης και βάσει του λογιστικού συστήματος μπορεί να γίνει η καθάριση των λογαριασμών. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη δεν υπάρχει καμία απόκληση με τον χρηματοδοτικό κανονισμό με τον οποίο η βάση του οποίου εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, τώρα, ε, η μέθοδος διόρθωσης ε, που έχει αποφασιστεί και από το ελεγκτικό συνέδριο στηρίζεται στην αναγνώριση της λειτουργίας του συστήματος. Όμως δεν μπορούμε άμεσα να δούμε ποιο είναι, ποιος είναι ο συγκεκριμένος δικαιούχος στον οποίο ε, οφείλεται η, η δυσλειτουργία. Εκεί εφαρμόζουμε λοιπόν αυτό το flat rate, δηλαδή αυτό το καταποκοπή διορθωτικό ποσό ε, και καλούμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ε, την συμμεριζόμενη διαχείριση επιτόπου. Επίσης, είχα πει προηγουμένως ότι αυτό το ποσό flat rate correction αναφέρεται ε, και στο δείγμα που έχουμε και στους ελέγχους που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Προτείναμε λοιπόν στα κράτη-μέλη τα οποία είχαν μπει στη διαδικασία flat rate correction ε, να ε, προσελθούν με περισσότερους ελέγχους επιτόπου και αν βάσει του αποτελέσματος ελέγχων που γίνονται επιτόπου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τότε μπορούμε να αποσύρουμε τις ε, παρατηρήσεις αυτές ε, μετά από συζήτηση και με τα κράτη-μέλη. Είναι όμως πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την δημοσίευση των δικαιούχων να πω μάλλον επίσης ότι για καταστάσεις όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία διαπιστώνουμε ότι το 2007 ήταν η, η πρώτη χρονιά που χρησιμοποίησαν οι χώρες αυτές αυτό το σύστημα. Στις επόμενες χρονιές, 2008-2009, ε, ε, είδαμε μία μείωση των ε, μια μείωση του λάθους και μια αύξηση των ελέγχων, πράγμα που σημαίνει ότι η τάση είναι πτωτική. Και βεβαίως και στο μέλλον θα πρέπει να διασφαλίσουμε περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού λάθους και βεβαίως να λάβουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε να προστατέψουμε τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μέσω των διορθώσεων. Τώρα το ζήτημα της δημοσιοποίησης των δικαιούχων και το θέμα της διαφάνειας. Το ε, δικαστήριο δεν αμφισβητεί την αρχή της διαφάνειας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ε, καλύψουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Η διαφάνεια υπάρχει και θέλουμε να τη διατηρήσουμε όμως με τον κανονισμό που ορίζει τις προϋποθέσεις ε, που θα πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη στη δημοσιοποίηση των ε, ονομάτων των δικαιούχων ε, θα πρέπει να καταλήγει σε καλύτερη προστασία των φυσικών προσώπων. Εγώ νομίζω ότι αφού πρόκειται για δημόσιο χρήμα, το οποίο δίνεται σε έναν ιδιώτη δικαιούχο, η διαδικασία διαφάνειας πρέπει να είναι σαφής και εν πάση περιπτώσει δεν θίγει τα ιδιωτικά ε, συμφέροντα του εν λόγω δικαιούχου. Επομένως, εφαρμόζουμε την αρχή της διαφάνειας και εντωμεταξύ ζητούμε από τα κράτη-μέλη του επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα, μέχρι δηλαδή την επόμενη δημοσιοποίηση, να κάνουν μια διαφοροποίηση ανάμεσα ε, στα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα. Να κάνουν λοιπόν το διαχωρισμό αυτό έτσι ώστε και την επόμενη χρονιά να μπορέσουμε τουλάχιστον να συνεχίσουμε τη δημοσιοποίηση για τα νομικά πρόσωπα και μετά να υπάρξει και περαιτέρω που αποσαφήνιση τις νομοθεσία για τα ιδιωτικά όσον αφορά τους ελέγχους επιτόπου για τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν λιγότερα προβλήματα, αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι ότι ε, στις περιοχές που συστηματικά έχουν χαμηλό ποσοστό λάθους και για να μειώσουμε ε, το διαχειριστικό κόστος ε, προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει μειωμένο ποσοστό ελέγχων γιατί τα προβλήματα που εμφανίζονται επί τόπου είναι ελάχιστα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα υπάρξει επαγρύπνηση και εποπτεία του συστήματος. Απλώς θα μειωθεί το ποσοστό του δείγματος εάν το ποσοστό λάθος είναι 0,02-0,03%. Ε, το ποσοστό ασφάλματος δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο ε, λειτουργεί και επομένως ε, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με το ίδιο δείγμα. Φυσικά για περιπτώσεις όπως της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας θα συνεχίσουμε με τα δείγματα τα κανονικά. το σύστημα, μέσα από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών των οργανισμών πληρωμής μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Το να έχουμε ένα help desk στην Κομισιόν, το να έχουμε ένα γραφείο στην Κομισιόν που θα, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορεί να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να λύσεις προβλήματα επιτόπου καθισμένο σε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες το κάλλιστο αποτέλεσμα ε, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συναντήσεις ε, των οργανισμών πληρωμής ε, των κρατών μελών. Μία τέτοια συνάντηση γίνεται δύο φορές το χρόνο για την ώρα. Ευελπιστούμε ότι θα μπορούν να συναντιούνται με πιο συχνό ρυθμό έτσι ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βλέπουν οι μεν με ποιο τρόπο ερμηνεύουν οι δε τον κανονισμό, να ανταλλάσσουν στοιχεία ο τρόπος εφαρμογής ε, ενός κανόνα επιτόπου είναι πολύ σημαντικός, πολύ σημαντικότερο σε πάση περιπτώσει από την ίδρυση ενός help desk στην Κομισιόν. Συνέλεφος ε, Γκάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η δική μου ερώτηση σχετίζεται με τα επιχειρήματα του εισηγητή μας που ακούστηκαν χθε, ο οποίος επεσήμανε ότι θα έπρεπε για να είμαι προσεκτικός το λέω αργά αργά, ε, σε κράτη για τα οποία γνωρίζουμε ότι κάπως τακτικά παραβιάζουν τους κανόνες, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να αναλυφθούν άμεσα μέτρα. Σας εύχομαι λοιπόν κύριε Επίτροπε κάθε επιτυχία ως προς την ε, μείωση του ποσοστού σφάλματος και εγώ προσωπικώς έχω δηλώσει ότι με ενδιαφέρει όπως και τη συνάδελφο Γκρέσλε να έχουμε ως το δυνατόν χαμηλό ποσοστό ε, σφάλματος και συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε πίσω ότι το 2 ή το 2 και 2,1-2,2% δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε στα κράτη αυτά τα οποία έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματος ε, να βοηθήσουμε με, με την απλούστευση των κανόνων έτσι ώστε να μην χρειάζεται να χάνουν χρόνο επαναλαμβάνοντας τις ε, ε επαληθεύσεις οποίες ανέφερε η κυρία Γκρέσλε νωρίτερα ε, και από την άλλη θα πρέπει να δούμε διαφορετικό μάτι εκείνους οι οποίοι βρίσκονται τακτικά στο κόκκινο, για να μην πω βαθύ κόκκινο. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή όμω έχει μια κάπω χαλαρή στάση. Λέει ότι ναι, το ξέρουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε κτλ. Ε, δεν αρκεί αυτό. Γιατί ασφαλώ στην ε, απόφαση, στο ψήφισμα για την απαλλαγή θα χρειαστεί να συζητήσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά τα τρία αυτά κράτη. Έτσι λοιπόν και μετά την ε, γραπτή μου ερώτηση σας παρακαλώ να μας πείτε τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα ώστε να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος και επίσης δεύτερη ερώτηση απευθυνώνει κυρίως προς το ελεκτικό συνέδριο σε μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής σε τις εκθέσεις Φερρυπίν θα υπάρξει μια πιο επακριβής ε, απαρίθμηση των περιπτώσεων και δι των κρατών που έχουν ε, διαπράξει το μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος. Απάντηση, ο κύριος Τσόλος. Για τα κράτη-μέλη που παρουσιάζουν τακτικά προβλήματα. Να σας πω. Το έχω πει πολλές φορές. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες πάντοτε παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες. Πολύ στενά. Στο τωρινό δημοσιονομικό κανονισμό δε έχουμε σαφέστατα κριτήρια βάσει των οποίων προχωρούμε προς το το μέτρο, δηλαδή την διακοπή των πληρωμών. Το είπα και θα το επαναλάβω, δεν διστάζω να διακόψω την καταβολή των ποσών ε, εφόσον αυτή είναι η μόνη λύση που μου μένει. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχω να σας πω ότι πριν από μερικές εβδομάδες μόνο απέστειλα επιστολή στους υπουργούς, τους δύο υπουργούς, ε, επισημένοντας ότι ε, καραδοκεί ο σχετικός κίνδυνος και ζητώντα του να βελτιώσουν πολύ σύντομα τι βάσει δεδομένων, διότι, παραλαμβάνω, πρόκειται αφενό μεν για το πρόβλημα του συστημικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου να μην λειτουργεί σωστά το σύστημα με τη βάση δεδομένων των αγροτεμαχίων, Αφενό, αφετέρου όμω υπάρχει και το πρόβλημα του πώ επαληθεύεται, πώ γίνεται δηλαδή ο επιτόπου έλεγχος ε, της λειτουργίας του συστήματος και εδώ έχουμε να κάνουμε προβλήματα κατάρτισης προσωπικού. Όμως η βάση δεδομένων πρέπει να είναι στη, αρχικά, καταρχήν, ορθή. Εδώ λοιπόν με το σύστημα εντοπισμού των αγροτεμαχιών, το LPAS, ε, έχουμε πρόβλημα στα δύο αυτά κράτη, Βουλγαρία, Ρουμάνια. Τώρα βλέπουμε ότι το, ξανα, ε, το αναθεωρούν, το βελτιώνουν, το επικαιροποιούν με τι νέε φωτογραφίσεις. Πρέπει να ολοκληρώσουν επίση τα δύο αυτά κράτη το σύστημα τη ε, μηχανογράφηση, τη ψηφιοποίηση καλύτερα αυτών των βάσεων δεδομένων για, τις, για τα αγροτεμάχια, έτσι ώστε στην προσεχή περίοδο κατάθεση αιτήσεων για ενίσχυση να μπορούν οι σχετικές υπηρεσίες να αξιοποιήσουν τα ε, βελτιωμένα στοιχεία. Είναι πολύ ξεκάθαρη λοιπόν η δράση την οποία πρέπει να αναλάβουν, οι συγκεκριμένε προθεσμίε και το τι έχουν να κάνουν και το τι θα ελέγξουμε όταν ελέγξουμε. Σας διαβεβαιώ, δεν πρόκειται να διστάσω ούτε δευτερόλεπτο να ε, επιβάλλω διακοπή των καταβολών εάν δω ότι δεν υπάρχει λύση. Παρατηρούμε όμω επίση το εξή, ότι από το καλοκαίρι που είδαμε του ελέγχου, από το Πάσχα καλύτερα πριν από τι τεράστιε διακοπέ, από την Άνοιξη μάλλον, ε, ε, υπάρχει μια πρόοδο και η απειλή αυτή ότι θα διακοπούν οι πληρωμέ φέρνει καρπού. Πέραν και εκπαραλύνουμε αυτή την απειλή για διακοπή πληρωμών, επιβάλλουμε και τι δημοσιονομικέ διορθώσει που ε, δώσαμε για 100 για το έτος 2007 στα δύο αυτά κράτη, ακριβώς γιατί υπήρχε κακή διαχείριση. Διόρθωση λοιπόν του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και το ίδιο γίνεται και το 2008. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε θα επιβληθεί η δημοσιονομική διόρθωση. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε του σύνεγγες. Το ίδιο για την Ελλάδα ήρθε η σχετική απειλή, γιατί τώρα, εφόσον επαληθεύθηκε, γιατί έγινε ο σχετικό έλεγχο του συστήματο, ότι η Ελλάδα έχει ένα σύστημα, ε, μια βάση δεδομένων αγροτεμαχίων αξιόπιστο, και έτσι ήρθε η απειλή, αλλά εάν οι έλεγχοι επιτόπου ε, διαπιστώνουν προβλήματα ή σφάλματα επιτόπου, γιατί σας είπα, ο το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε κακή ταυτοποίηση ε, αγροτεμαχίου από τον γεωργό στο ψηφιοποιημένο χάρτη ή μπορεί να οφείλεται και σε λάθος δήλωση του γεωργού ως προς το τι έχει πάνω στο αγροτεμαχιό του. Άρα εδώ χρειάζονται και καλύτερες τεχνικές φύσεως συμβουλές για τον γεωργό, για τον ε, ε, κτηνοτρόφο. Το έχουμε πει αυτό στα κρατημέλη ότι χρειάζονται καλύτερη υποστήριξη οι γεωργοί την ώρα που έρχονται να κάνουν τη δήλωση με μαχείου την ώρα που υποβάλλουν την αίτησή του. Και βέβαια πρέπει να βελτιώσουν τα κρατημέλη και του ελέγχου. Όμω αυτό το παρακολουθούμε κάθε χρόνο ε, πολύ προσεκτικά με αυτό το σύστημα του δημοσιονομικ... της δημοσιονομικής διορθώσεως. Άλλα κρατημέλη τώρα που ήδη έχουμε ε, βάλει στο στόχαστρο σημειώνουν τα τελευταία χρόνια ε, επανειλημμένα σφάλματα, διαδοχικά σφάλματα και πάλι ζητούμε πρόγραμμα δράσης και πάλι επαληθεύουμε ότι ε, βελτιώνεται το πρόβλημα και αν δεν βελτιωθεί αναλαμβάνουμε μέτρα με τελικά την επαπειλούμενη διακοπή των πληρωμών. Σε αυτό είμαι άτεγκτος. Ο, ο κύριος Κρατέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα του κυρίου Γκάγερ για το ποσοστό δημοσίευσης φαρμάτων ανακράτος μέλος. Η εύκολη απάντηση είναι αρνητική. Δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε κάτι τέτοιο για τους λόγους που σας παρουσίασα όταν απάντησα στον κύριο όταν μίλησα για τους ελέγχους. Δηλαδή, εμείς ε, κάνουμε δειγματοληψία για τα 27 κράτη-μέλη, όχι ανά κράτος μέλος. Επομένως εξετάζουμε το πράγματα στο σύνολο της κοινότητας και όντως προκύπτει κάθε χρονιά ότι ορισμένες πληρωμές έχουν γίνει σε ορισμένες χώρες και δεν ε, βρίσκονται στο δείγμα, γιατί το δείγμα επιλέγεται τυχαία επί του συνόλου των πληρωμών που έχουν γίνει στο σύνολο των 27 κρατών μελών. Δεν εξετάζουμε δείγμα αναχώρα ατομικά, ξεχωριστά. Επομένως δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τέτοιο είδος ποσοστού σφαλμάτων ανακράτος και δεν καλούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο από τη συνθήκη. Η συνθήκη μας, ζητεί, ε, μας ζητά να αποφανθούμε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σύνολό του. Βεβαίως ε, ενισχύουμε τους ελέγχους μας με το σύστημα χωρών υψηλού κινδύνου και παρακολουθούμε την κατάσταση για να δούμε τι γίνεται και μετά ε, τη πρώτη διαπίστωση, τη διαπίστωση ε, κάποιων πρώτων παρατηρήσεων. Και το ίδιο συνέβη και με τη Βουλγαρία και γι' αυτό σας έδωσα αυτά τα στοιχεία προηγουμένως. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα οποία συνέβησαν στη Βουλγαρία δεν συνιστούν σφάλμα. Παρόλα αυτά, φέτος, οι ίδιες οι βουλγαρικές αρχές παρακράτησαν τις πληρωμές, δηλαδή δέσμευσαν, διέκοψαν τις πληρωμές, δηλαδή υποψιάζονταν ε, σφάλμα. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να ενισχύουμε τον έλεγχο των ε, συστημάτων στις χώρες όπου ο κίνδυνος είναι υψηλότερο συγκριτικά με τις άλλες. Ενισχύουμε λοιπόν τα συστήματα ελέγχου και έτσι ε, εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς θα βελτιωθούν οι έλεγχοι στις εν λόγω χώρες. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε να πω και δύο λόγια για την παρέμβαση της κυρίας Γκρέσλε. Ως προς την εκαθάριση λογαριασμών έχει υποβληθεί η έκταση και θα, θα εξεταστεί λίγα συντόμως από την Επιτροπή σας. Το ελεγκτικό συνέδριο παραμένει διατηρεί ε, τις ε, διαπιστώσεις ε, που φαίνονται στην έκθεση αυτή. Επιμένουμε σε αυτές, θα το συζητήσουμε όμως εν ευθέτω χρόνο. Ο συνάδελφος από το ελεγκτικό συνέδριο. Συμφωνώ κύριε Πρόεδρε με αυτά που είπε ο συνηγητής, ο κύριος Κρετέν. Ως προς τον πρώτο πυλώνα για τον οποίο είμαι αρμόδιος θα έλεγα ότι, ότι χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις για να βελτιωθεί γενικότερα το σύστημα ελέγχου των συναλλαγών. Ως προς τα συστήματα ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων, δεν αποκλείστηκαν πάντοτε μη επιλέξιμα σφάλματα ως προς τους ελέγχους επιτόπου. Πολύ συχνά δεν έχει εφαρμοστεί σωστά η αρχή της μη ανεκτικότητας. Και ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση δεν έχει προσδιορίσει το κράτος μέλος αυτό το οποίο ε, χρειάζεται και πρέπει να τηρείται ώστε όντως να χαρακτηριστεί η έκταση ότι διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Ε, νωρίτερα έγινε λόγος ε, για επιληρωμές που έχουν γίνει για τη βελτίωση της γεωργικής δραστηριότητας. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση αυτή έγιναν πολλοί έλεγχοι και στον έλεγχο πριν από δύο εβδομάδες έγιναν δεκτά μόνο τα 400 εκτάρια από τα 500. Και για το 2009 οι εθνικές αρχές δεν πλήρωσαν τίποτα. Δεν έχει δηλαδή εκταμιευτεί ε, κάποιο ποσό για το 2009-2010. Είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση και μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία ε, στον εισηγητή αν τα χρειάζεται, στην εισηγήτρια. Στις συστάσεις μας λέμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν κανόνες ως προς τις πληρωμές και θα πρέπει ε, για τα βοσκοτόπια να έχει σε επίπεδο επιτροπής να τεθούν ετήσιες προϋποθέσεις, ελάχιστες μήνυμου προϋποθέσεις ετήσιες για να ε, χαρακτηριστούν ως τέτοιες οι εκτάσεις αυτές. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, μια μεταρρύθμιση η οποία ε, όντως είναι πρόοδος. Ο Επίτροπος, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το θέμα του δείγματος ανακράτος μέλους και ποσοστό ε, σφάλματος ανάκρατος μέλος. Όλα αυτά είναι στοιχεία που υπάρχουν στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την οποία υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής, ε, με βάση αυτά τα οποία υποβάλλουν σε εμάς οι εθνικές αρχές, τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει. Προτίθεται να ζητήσει από τα κράτη-μέλη, από τους οργανισμούς πιστοποίησης, να πιστοποιήσουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία με βάση αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα ανά κράτος μέλος και ανά ε, μέτρο αν θέλετε. Και με βάση αυτό το αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα ε, τα στοιχεία υποβάλλονται από τους οργανισμούς πληρωμών και έτσι μπορούμε να δημοσιεύουμε ε, σαφή και αντιπροσωπευτικά στοιχεία και πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Ε, μπορούμε μετά ως Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τα αναλύσει και το Ελεκτικό Συνέδριο επίσης. Δεν θέλω να επιμείνω στις ε, ξεχωριστές συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα επανέλθω όμως γιατί ο κύριος Κατά υπογράμμισε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι η Βουλγαρία ανέστηλε, διέκοψε τις πληρωμές ε, για την περίπτωση αυτή για το παράδειγμα που αναφέρθηκε. Ναι, το απέσυρε η Βουλγαρία γιατί ε, βάσει των διαπιστώσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Όταν το ελεκτικό συνέδριο κάνει συγκεκριμένε διαπιστώσει, ένα κράτο μέλο δεν μπορεί παρά να τι λάβει υπόψη του. Επιμένω όμω εγώ στου ελέγχου που κάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, στι φωτογραφίε που λαμβάνουμε, στη βάση των δεδομένων, ε, στου σαφεί ορισμού για το τι εστί επιλέξιμο αγροτεμάχιο, και αν γινόταν αυτή η τριμερή σύσκεψη ε, ίσως θα ήταν την καλύτερη κατάσταση. Το γεγονός ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, ε, συσκέπτεται με τις εθνικές αρχές και μετά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δεν αποτελεί τριμερή διαδικασία. Ίσως θα πρέπει να καθίσουμε στο, γύρω από ένα τραπέζι και τα τρία μέλη τα τρία μέρη για να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Εμεί πάντοτε είμαστε ανοιχτοί. Όταν δεν υπάρχουν επιχειρήματα το αναγνωρίζουμε αυτό. Και άλλωστε αυτό έχει συμβεί για συγκεκριμένε παρατηρήσει του ελεκτικού συνεδρίου. Ε, σε κάθε περίπτωση το ελεκτικό συνέδριο μπορεί να βασιστεί στο πνεύμα συνεργασίας, στο ανοιχτό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκρινιστεί η κατάσταση. Όμως ως Επιτροπή εφαρμόζουμε και τους κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολύ σύντομα μία ερώτηση σχετικά με την απλούστευση της ΚΑΠΑ. Το Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες ενέκρινε την έκθεση ΣΦΟΡΠ ε, για την απλούστευση και εκεί γινόταν αναφορά ειδική στις πληρωμές ε, πληρωμές οι οποίες δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει και το Κοινοβούλιο ε, διεπίστωσε ότι δεν ε, υπήρχαν περιπτώσεις ε, για τις ε, οποίες να πιέστηκαν μονόμενα άτομα να επιστρέψουν τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Κυρίως ανεπρόκειτο για λάθη άλλων. Ξέρουμε στην Πολωνία λάθη που έγιναν από το κράτος. Στην Πολωνία δυστυχώς υπάρχουν γεωργοί ε, οι οποίοι, δεν, ε, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν χρήματα ε, κυρίως γιατί δεν καλύπτουν κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Και μία άλλη ερώτηση που μου έχουν θέσει οι ψηφοφόροι μου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σύζυγος του ε, ε, γεωργού έχει μια δικιά της εκμετάλλευση. Ε, εκεί φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να πιστούν οι σύζυγοι να έχουν από κοινού κάποια αίτηση, δηλαδή να παίρνουν τα χρήματα από κοινού. Ε, ποια είναι η άποψή σας, θα πρέπει να παραμείνει ο κάθε γεωργός ε, να πληρώνεται για το αγροτεμάτιχιό του, για την εκμετάλλευσή του ή θα πρέπει σε περίπτωση συζύγων οι δύο σύζυγοι ε, να έχουν κοινή αντιμετώπιση. Θα ήθελα απάντηση γιατί απασχολεί πολύ αυτό τους ψηφοφόρους μου. Όσον αφορά την απλούστευση, απαντάει ο Επίτροπος, ε, χαίρομαι που θέτετε το θέμα αυτό, γιατί ε, έρχομαι και στην Επιτροπή Γεωργίας και ακούω ε, τους προβληματισμούς σας και βεβαίως ρόλος μου μεταξύ άλλων είναι να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και βεβαίως πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την κόκκινη γραμμή της απλούστευσης, δηλαδή να μην υπεραπλουστεύσουμε τόσο ώστε να αποδυναμώσουμε τελικά τη διαδικασία. Αυτό που θέλουμε είναι να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες της Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, οι διαδικασίες που εφαρμόζουν επιτόπου ε, τα κράτη-μέλη, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και αυτού του είδους η έλεγχη, η δεύτερη έλεγχη των κρατών μελών, αυτοί διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Πρέπει να δούμε λοιπόν την απλούστευση στο σύνολό της και ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης ε, που του πρέπει. Όσον αφορά τώρα την επιστροφή. Όταν, το κράτ, όταν ο δικαιούχος ε, ευθύνεται θα πρέπει το, ο δικαιούχος να επιστρέψει τα χρήματα. Εάν όμως ευθύνονται τα κράτη-μέλη, επιστρέφουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν ε, διαδικασίες διόρθωσης που αφορούν τα κράτη-μέλη και σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς πληρώνουν τα κράτη-μέλη. Όταν όμως ε, πρέπει να γίνει διόρθωση από πλευράς του δικαιούχου, τότε ή θα πληρώσει ο δικαιούχος ή θα χρεωθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Σε περίπτωση συζύγων δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα αυτό. Ούτε απαγορευτική, ε, δηλαδή να μην ενωθούν οι σύζυγοι, ούτε ε, ε, υποχρεωτική προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Τώρα, το τι κάνει η Πολωνία είναι δικό της θέμα. Ενδεχομένως, λοιπόν, αυτή η τάση στην Πολωνία, οι δύο σύζυγοι, έστω και αν έχουν χωριστές εκμεταλλεύσεις, να ζητούν από κοινού ε, τα κονδύλια, είναι προφανώς ε, ε, πολωνικό ζήτημα. μία τελευταία δήλωση του κυρίου Χατζημαρκάκη, του εισηγητού. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι εκφράζω και τους συναδέλφους λέγοντας ότι διαπιστώνω πως γνωρίζετε πολύ καλά τον τομέα σας. Δεν ήταν τόσο καλή η προκάτοχή σας στη θέση του Επιτρόπου, σας το λέω αυτό, με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπό τους. Πρέπει να το πούμε λοιπόν. Από την άλλη είναι ξεκάθαρο, όταν καλής ξέρει καλά τη δουλειά του, μπορεί κανείς να είναι και πιο απαιτητικό και να, να τον καλεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί από όλες τις πολιτικές ομάδες όπως και εγώ έχουμε κάθε σεβασμό για τα όσα μας είπατε σήμερα εδώ. Πιστεύουμε ότι είστε ο σωστός επίτροπος, ο επίτροπος εκείνος ο οποίος μπορεί πράγματι να φέρει πέρα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρώτο θέμα λοιπόν, απλούστευση το ελεγκτικό συνέδριο μας με τον κύριο Νίσελε αλλά και τον κύριο Κρετέ, αλλά και εσείς κύριε Τσόλος είπατε ότι θα υπάρξει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της απλούστευσης. Πολύ καλά. Από εσάς από το ελεγκτικό συνέδριο ακούσαμε ξεκάθαρες προτάσεις για την υπαγωγή σε όρους και όχι μόνο. Ε, ένα πρόγραμμα δράσεως λοιπόν το οποίο πιστεύουμε ότι μπορείτε να αναλάβετε και για το οποίο μπορούμε να περιμένουμε ε, σαφείς ορισμούς μέχρι την Άνοιξη. Αναφέρθηκε αυτό το θέμα ήδη και είμαι αισιόδοξο ότι θα το ολοκληρώσετε. Επίσης μιλήσατε για το όλο πλέγμα των ποινών, απειλών και διακοπών πληρωμών. Περίπλοκο πλέγμα, σημαντικό πλέγμα πάνω απ' όλα. Πρώτον, κυρώσεις. Για την ανάκτηση των κονδυλίων είπατε ότι βελτιούται, ναι, αλλά έχουμε φτάσει μόνο στο μισό γιατί το υπόλοιπο μισό με το σύστημα που έχουμε παραμένει στα χέρια εκείνου που αχρεωσίτως το εισέπραξε. Έτσι λοιπόν οι απειλές ω δεύτερο μέσον καλέ είναι, δεν επαρκούν όμω πολλέ φορέ και έτσι θα πρέπει να προχωρούμε και στη διακοπή και ακόμη στην πάυση, εάν χρειαστεί. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα σε μια παρατήρηση του συναδέλφου Οντί, ο οποίο είπε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στι εθνικέ δηλώσει. Εγώ με τον κύριο Μίλτερ και τον κύριο Τέρι Γουίν, αν δεν με το 2004 ήταν η πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα αυτό, διεκδικήσαμε δηλαδή τέτοιου είδους ε, δηλώσεις από, τα, από τις κυβερνήσεις, από τα κράτη, με την απαλλαγή εκείνη και δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε να υπάρξει αυτό το σύστημα και νομίζω ότι θα ήταν καλό, όπως είπε και ο κύριος Σοντή, να εμπλακούν και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια στην υπόθεση αυτή. Όπω είπε και ο κύριο Κρέτα νωρίτερα. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσεται τη ευθύνη ο Υπουργό των Οικονομικών τη κάθε χώρα, εκείνο δηλαδή ο οποίο έχει να επιτελέσει το σχετικό έργο. Και νομίζω ότι μπορούμε και μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου για άλλη μια φορά να αποστείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου ω Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να διεκδικήσουμε να μιλήσουμε με το ΕΚΟΦΗΝ. Στο ΕΚΟΦΗΝ έχουμε υπουργού των οικονομικών οι οποίοι ναι ασχολούνται με το ευρώ και πολλά άλλα σημαντικά θέματα αλλά καλό θα ήταν να ασχολούνται πότε πότε και με την διοίκηση των υπουργείων του, δηλαδή τη διαχείριση τη δουλειά που πραγματικά έχουν αναλάβει. Τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν προκαλέσει και τα μεγάλα προβλήματα τώρα στο ευρώ όπω η Ελλάδα πρέπει να κληθούν σε, περισσότερη, σε περισσότερο πειθαρχημένη συμπεριφορά. Μεγάλο κομμάτι του προπολογισμού που βγήκε από τα δικά σα τα ταμεία πήγε στην Ελλάδα κατά τρόπο που δεν ήταν σύμφωνο με του κανόνε και άρα χρειάζεται περισσότερη ευρωπιθαρχία. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με το ΕΚΟΦΗΝ και, εν πάση περιπτώσει, να ασκήσουμε πίεση για να καταστούν σαφεί οι θέσει μα. Οι δηλώσει λοιπόν από την διοίκηση των κρατών είναι πολύ σημαντικό μέσο το οποίο δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε, το οποίο θα διεκδικούμε διαρκώ. Πάντω ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρουσία σα εδώ και γενικά για τη δουλειά σας και ενώπιον του Συμβουλίου, νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο τα παραδείγματα, αυτά τα καλά παραδείγματα, έτσι ώστε να διαδοθούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζημαρκάκη, ευχαριστούμε πολύ και τον Επίτροπο Τσιόλος γιατί ήταν μαζί μας για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχαμε ε, αρχικά προτείνει. Περανάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, σημείο 8 η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου 5 κάθετο 2010 εφαρμογή τη προσέγγιση Λίντρια για την ανάπτυξη τη υπαίθρου δίνω το λόγο στον κύριο Ντέρεκ Βόγκαν, τον εισηγητή μα. Yeah, thank you, Chair. was just pausing a second. Αρχίστε, γιατί αν δεν αρχίσετε να μιλάτε δεν θα φύγει κανείς από την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή του. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε και ξαναευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Ιδίω ε, δε και τον κύριο Λαζάρου, το νερό μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που ήταν υπεύθυνο για αυτήν την συγκεκριμένη έκθεση. Πρέπει να πω εξ ε, ότι ε, ε, είμαι απολύτως υπέρ αυτής της νέας προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε μονάχα να ενισχύσουμε την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες παρόλο που κατανοώ το σημείο που αναφέρει το συνέδριο ότι δεν είναι πάντα εφικτή η προσωμέτρηση αυτών και η αποτίμηση μάλλον αυτών ε, των, της προστιθέμενης αξίας τέτοιων ε, πρωτοβουλειών. Ε, και βεβαίως το στοιχείο αυτό θα μπει ενδεχομένως και στην uh, και στην απαλλαγή. Το 2000 είχε γίνει το, η προηγούμενη έκθεση για το θέμα αυτό και ενδεχομένως ε, γι' αυτό ε, αιτιολογείται και η κρισιμότητα της έκθεσης ε, του συνεδρίου. με ενδιαφέρουν περισσότερο οι προτάσεις 3, 4, 5 και 6 του ελεγκτικού συνεδρίου και επίσης όσον αφορά τη σύσταση 1 και 2 έχω να κάνω κάποια σχόλια. Για την σύσταση 1 συμμερίζομαι τα περισσότερα περισσότερα στοιχεία που αναφέρονται Δηλαδή, εάν ένα έργο έχει ολοκληρωθεί, τότε ε, δεν θα πρέπει να πάρει χρήματα από το Λίτερ. Όσον αφορά την ε, ευελιξία, ε, εάν, ας πούμε, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει και θέλει να μεγαλώσει, τότε, εάν συμπληρώνονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι μπορούν να ζητήσουν και επιπλέον χρηματοδότηση χρηματοδότηση και επομένως αυτή η ευελιξία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα. Όσον αφορά την δεύτερη σύσταση, αναφέρει το συνέδριο ότι ε, θα πρέπει να απουσιάζουν, δεν θα πρέπει να είναι παρόντα δηλαδή τα μέλη των ε, ομάδων τοπικής δράσης από τις ε, συζητήσεις, εκτιμήσεις ή αποφάσεις για το, θέμα, και για το έργο και το θέμα θα πρέπει να παραπέμπεται στη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ε, όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι ποτέ παρόντα τα μέλη. Όμως θα συμφωνήσω με, με το συνέδριο ότι οπωσδήποτε θα πρέπει εξ αρχής να γίνεται δήλωση ενδιαφέροντος και επίσης ότι τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων θα πρέπει να καταγράφονται και να δημοσιοποιούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιο τρόπο να διευρύνουμε ε, τα μέλη των οργανισμών τοπικής ε, δράσης έτσι ώστε πραγματικά να ενισχυθεί η συμμετοχή τη τοπικής κοινωνία. Ε, Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, να το ευχαριστήσω ιδιαιτέρω για τις ε, συστάσεις ε, οι οποίες θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικοδομητικέ, ακόμα και οι συστάσεις από των οποίων έχω κάποιες ενστάσεις θεωρώ ότι είναι πολύ αποτελεσματικές για τις ΟΔΤ επίσης ε, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει χρηστή διαχείριση αλλά φυσικά και να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε ε, τα ωφέλη, να είναι πολλά για τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λαζάρου από το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 5-20-10 συλλογική προσέγγιση στην ανάπτυξη πέθρου. Επιτρέψτε μου όμως να πω, ξεκινώντας, ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα το να είμαι στη θέση να παρουσιάσω ενώπιον τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού την πρώτη μου έκθεση και μάλιστα τόσο νωρί από την ε, μετά την, ε, τόσο γρήγορα μετά την ε, προηγούμενη μου παρουσία στο Σεπτέμβριο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου στις 2 Νοεμβρίου. Η έκθεση λοιπόν αυτή, όπως έχει σχεδιαστεί, έχει συνταχθεί υπό τον κύριο Καζαμία, ο οποίος ήταν ο προκάτοχός μου και ο οποίος έχει βέβαια αναλάβει όλη τη δουλειά. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά και όλη την υποστήριξη που μας προσέφερε. Εκπροσωπεί την Κύπρο, εκπροσώπησε μάλλον την Κύπρο στο Ελεκτικό Συνέδριο τα τελευταία έξι χρόνια. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Βον για την επακριβή καταγραφή της ε, έκθεσης και για τις συστάσεις του. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω επίσης για τις συστάσεις του, ιδιαίτερα για αυτήν την οποία έχει καταγράψει ως προς την ενίσχυση της προσέγγισης ε, προσθέμενης αξίας και της ε, χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης, διαχείρισης των σχεδίων των προγραμμάτων leader. Ιδιαίτερα λοιπόν οι ομάδες τοπικής δράσης είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν προσθέμενη αξία σε μία ε, προσέγγιση των κάτω προς τα άνω με μέτρα που έχουν προσδιοριστεί σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης οι ομάδες τοπικής δράσης όπως ήταν προβλεπόμενο, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τους εθνικούς στόχους, δεδομένου ότι η διαχείριση από τις αρχές δεν απαιτούσαν από αυτές λογοδοσία για τις επιδόσεις τους στους τομείς αυτούς. Πλην όμως το ε, έγγραφο εργασίας δεν υποστηρίζει, ε, δεν αποδεικνύει πλήρως τη χρησιμότητα των δύο συστάσεων, Για το ελεκτικό συνέδριο πιστεύει ότι αυτές οι δύο συστάσει που στόχο έχουν να αποφύγουν την ε, σύγκρουση συμφερόντων και να προστατεύσουν τα ε, ευρωπαϊκά χρήματα, τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό πρέπει να υποστηριχθούν. Έτσι λοιπόν, μετά την άρνηση της απαλλαγής ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει πάρει την πρωτοκαθεδρία στην ε, καταπολέμηση κάθε μορφής ε, συγκρούσεων συμφυρόντων, που άλλωστε περιλαμβάνονται και στο δημοσιονομικό κανονισμό στο άρθρο 52, ακριβώς για να αποτρέπονται τέτοιους καταστάσεις. Παρά την απαγόρευση το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι είναι εκτεταμένες περιπτώσεις των συγκρούσεων συμφερόντων και ειδικότερα ο κίνδυνος να λαμβάνουν τοπικοί παράγοντες τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των τοπικών προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν εδώ ε, ούτε επιλύονται τα προβλήματα τα οποία έχει επισημάνει το συνέδριο, ούτε και ε, επαρκούν τα μέσα του δημοσιονομικού κανονισμού για να αποτρέψουν δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, δεν πρόκειται για οικογενειακή κοινωνικούς δεσμούς, συναισθηματικούς, οικονομικούς ή πολιτικούς. Πολιτικά συμφέροντα. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για ένα ερώτημα ακαδημαϊκό, γιατί οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να έχουν πολύ σημαντική ε, επίπτωση ως προς τη λειτουργία του προγράμματος. Βλέπουμε λοιπόν ε, project, σχέδια τα οποία έχουν προαχθεί από τους ε, παράγοντες των τοπικών ομάδων δράσης και ιδιαίτερα στο παράδειγμα της Ιρλανδίας που επισημαίνει η έκθεση της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου φαίνεται ότι μπορεί η ομάδα δράσης να προσαρμοστεί στους κανόνες και τους προδιαγραφές του κανονισμού χωρίς να περιορίσει τις αστριότητές της. Η Επιτροπή απαντώντας στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να αποτρέπονται ή συγκρούσει συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια καλέσε τα κράτη-μέλη και μέσω των εκπροσώπων τους να παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή την κατάσταση ώστε να μην επιτρέπουν ανάπτυξη συγκρούσεων συμφερόντων που θα μπορούσαν να αμαυρώσουν την προσέγγιση leader Και γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω και την σύσταση του εισηγητού ε, για την προσέγγιση που σημαίνει ε, όρους υλοποίηση χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η δεύτερη σύσταση που δεν έτυχε πλήρω υποστήριξη ήταν αυτή που είχε να κάνει με ενίσχυση σχεδίων, με χορήγηση των κονδυλίων σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ένα από τα καθήκοντά μα είναι να βλέπουμε, να εντοπίσουμε πού μπορεί να βελτιωθεί ε, η διαχείριση των ε, δημόσιων κονδυλίων, πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό σε περιόδου δεινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση για πολλά κράτη-μέλη και πολλού ιδιαίτερα από του πολίτε των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην έκθεσή μας ότι υπάρχει ανάγκη για απερίφραστους και σαφείς κανόνες. Ε, χρηματοδότηση δεν μπορεί να δίνεται σε σχέδια που έχουν ξεκινήσει πριν ληφθεί η απόφαση για ε, μια χρηματοδότηση leader. Και επίσης θα πρέπει εάν δόθη εσφαλμένη απάντηση, απόφαση ή υπόσχεση για χρηματοδότηση ενός σχεδίου που έχει ήδη ξεκινήσει, εάν υπήρξε ε, συγκεκριμένη κατάχρηση, εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να διακόπτεται η χρηματοδότηση. Το να χορηγηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις τα κονδύλια είναι πολύ κακή δημοσιονομική διαχείριση. Όπω αναφέρεται λοιπόν από τον εισηγητή στην έκθεσή του, ένα σχέδιο το οποίο ήδη υφίσταται και είναι σημαντικό για την τοπική στρατηγική μπορεί να επεκταθεί χάρη στα κονδύλια Λίντερ και τότε μπορεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του σχεδίου, αλλά με προπόθεση ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται πριν από την επέκταση, πριν να ξεκινήσει η επέκταση του σχεδίου. Και εν τέλει, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι μέλη τη Επιτροπή σα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα προβλήματα τα οποία περιγράφω δεν έχουν ακόμη επιληθεί. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τελευταία έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το Λίντερ και δεν έχουν ακόμη επιληθεί τα προβλήματα αυτά. Και έτσι είναι καθήκον μου να υπογραμμίσω τη σημασία που αποδίδουμε στην σαφή υποστήριξη από την Επιτροπή σα, τη διαδικασία για την απαλλαγή, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό το Λίντερ, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι συγκρούσεω συμφερόντων, οι οποίε οι οποίες συγκρούσει συμφερόντων παραβλάπτουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και που τελικά δεν βοηθούν καθόλου στην ανάπτυξη Πέθρο, Ευχαριστώ πολύ. Ε, Θέλει να πάρει το λόγο κάποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω εσάς αλλά και τον κύριο Βόν και τον κύριο Λαζάρου και του, τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου διότι μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ ενώπιόν σας και να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το εργαλείο που είναι τόσο σημαντικό, το leader, για την πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και τον εισηγητή για τις συστάσεις τους. Βάσει όσων άκουσα, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ε, το πόσο μεγάλης εκτίμησης χαίρει η μέθοδος leader ε, διότι η προσέγγιση που ακολουθεί είναι από κάτω προς τα πάνω και καλεί τους τοπικούς φορείς να συμμετάσχουν. Ε, γίνεται κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη και πάρα πολλά καθήκοντα αναθέτονται σε τοπικό επίπεδο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του leader είναι αυτά που συγκροτούν και την προστιθέμενή του αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό του Λίντερ, σεβόμενη πάντοτε τη βασική αρχή της χρηστής ε, οικονομικής διαχείρισης. Υπό αυτή την έννοια λαμβάνουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Να είστε βέβαιοι ότι ήδη τις εφαρμόζουμε, τις υλοποιούμε, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ε, για τη διάρκεια, για το υπόλοιπο της ε, τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω ε, το ότι το leader δεν ε, συνιστά μια στατική έννοια. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Καταρχάς επρόκειτο για μια κοινοτική πρωτοβουλία. Μετά άλλαξε, έγινε το Leader Plus, Leader Sin και τώρα έγινε ο άξονας υπαριθμών 4 της πολιτικής μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η προσέγγιση που ακολουθούμε δηλαδή είναι μια προσέγγιση ε, ζωντανή που εξελίσσεται. Έχουμε ε, περίπου 2.000 ε, ομάδες, τοπικές ομάδες δράσης στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη σωστή πλαισίωση της υλοποίησης του Λίντερ και η προσπάθειά μας ε, αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Καταρχάς στο κανονιστικό επίπεδο. Διευκρινίζουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται. Κατά δεύτερο λόγο, ε, δίνουμε πρακτικούς προσανατολισμούς, ε, κατευθυντήριες γραμμές στις εθνικές αρχές για να εγκρίνουν τα προγράμματα που υποβάλλονται. Και στη συνέχεια με τις συστάσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους ε, προβαίνουμε στην εφαρμογή των ε, οικονομικών διορθώσεων. Και τέλος, εδώ και δύο χρόνια έχουμε μία μόνιμη συνοδεία, αν θέλετε, ε, παρακολούθηση εκ του σύνδεκης ε, στο πλαίσιο του δικτύου για τις ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, λειτουργεί μια υποεπιτροπή leader με βάση τη δουλειά των focus group. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του δικτύου και των focus group θα καταρτήσουμε μια έκθεση που θα αναλύει αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και θα αναλύει αυτό το καινοτόμο χαρακτήρα ε, της έννοιας του leader και θα αναλύει και την συνεργασία που γίνεται. Ε, πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη η έκθεση αυτή και θα είστε σε θέση να την ε, διαβάσετε. Επιθυμούμε καλύτερο διαχωρισμό των διαφόρων καθηκόντων των διαφόρων αρχών ε, διαχείρισης και διοίκησης και μεταξύ των κεντρικών αρχών και των τοπικών ομάδων δράσης, των ΛΑΓ ώστε να υλοποιούνται όλα αυτά τα ενοποιημένα προγράμματα. Και για να μην ε, μπω σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ελεκτικό Συνέδριο εργάζεται, ε, έχει αναλάβει ήδη αυτές τις δεσμεύσεις, εγκρίνοντας τα προγράμματα ή εγκρίνοντας τις τροποποιήσεις στα προγράμματα. Σας καλώ να διαβάσετε το σημείο 91 της έκθεσης. Εκεί υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες του κανονισμού 1974. για την έγκριση και την τροποποίηση, την έγκριση της τροποποίησης των προγραμμάτων. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε εμείς και ε, είναι και η απάντησή μας στις συστάσεις 3 και 5 ε, του ελεκτικού συνεδρίου, έτσι όπως ε, απεικονίζονται στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω αυτό το οποίο έχει να κάνει με την αξιολόγηση του Leader Plus. Θα έχουμε ε, αργότερα αυτή τη χρονιά μια έκθεση ex post, εκ των προτέρων, έκθεση αξιολόγησης του Leader Plus, εκ των υστέρων με συγχωρείτε, ex post, και ε, αυτή τη δουλειά θα την κάνουμε και στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Επιτροπής για τα θέματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Δηλαδή θα αναλύσουμε και την προοπτική του δικτύου αλλά θα λειτουργήσουμε και πολύ εστιασμένα σε συνεργασία με τις διαχειριστικές επιτροπές. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου ε, εκφράζοντας τη συμφωνία μου με αυτό το οποίο ε, λέγεται στην σύσταση, αναφέρεται στη σύσταση υπαριθμών 1 του ελεκτικού συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με αυτό. Όντως, ε, με την ευθυγράμμιση που γίνεται βάσει ε, της συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση και με τον κανονισμό 1698, τροποποιείται λοιπόν ο βασικός κανονισμός, ώστε για να διευκρι... ώστε να διευκρινιστεί καλύτερη... καλύτερα η κατάσταση. Ε, το ΦΕΑΝΤΕΡ να στηρίζει μετά την υποβολή του αιτήματο. Όλα αυτά ε, τα εξετάζει το Συμβούλιο, έχουν πάει στο Συμβούλιο ήδη αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στη σύσταση παριθμών 1 του ελεκτικού συνεδρίου. Ως προς τη σύγκρουση ε, συμφερόντων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε για να ε, έχουμε σωστή διαχείριση και μέγιστη προστιθέμενη αξία. Εξού και τροποποιούμε τον κανονισμό που προβλέπει τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες. Και ε, αυτό ήδη θα παρουσιαστεί στη Διαχειριστική Επιτροπή ή Δεκέμβριο-Ιανουάριο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για να έχουμε διπλή απαρτία, έτσι το ονομάζουμε. Δηλαδή, οι αποφάσεις και οι ψηφοφορίες να μην γίνονται χωρίς να τηρείται το ελάχιστο του 50% της συμμετοχής 50% από την πλευρά των τοπικών ομάδων δράσης, των τοπικών φορέων. ώστε να υπάρξει σωστή διαχείριση. Αυτό φαίνεται και με τον οδηγό που θα υπάρξει και θα συζητηθεί στην ίδια Διαχειριστική Επιτροπή ήδη το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Τέλος, ή μάλλον να σχολιάσω ε, ένα άλλο σημείο της έκθεσης με, τον με το οποίο είμαστε απόλυτο σύμφωνοι. Η τοπική στρατηγική εκάστοτε θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία, να είναι ποιοτική και να συνοδεύεται από όσο το δυνατόν πιο μετρήσιμους στόχους. Ε, σε αυτό θα βοηθήσει ο οδηγός διότι θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες διευκρινήσεις για να βελτιωθεί η ποιότητα της στρατηγικής. Επομένως και σε αυτό είναι χρήσιμος ο οδηγός. Τέλος, ως προς τα σχόλια του εισηγητή ε, για ε, τους τοπικούς φορείς και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα ε, τις ε, κατατόπους δυνατότητες. Έχουμε ένα μόνιμο διάλογο ξεκινήσει με τα δίκτυα και αυτό είναι μέλημά μας ε, στη χάραξη των αρχών για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα, ως προς τη διαφάνεια, στον οδηγό θα υπάρχουν σίγουρα οι απαραίτητες διευκρινήσεις για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, δημοσίευση των πεπραγμένων, ε, μεταξύ άλλων. Κύριε Πρόεδρε, ε, Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τελειοποιήσει την προσέγγιση Leader, μια προσέγγιση η οποία είναι κλειδί ώστε η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου πράγματι να ικανοποιεί τις ανάγκες ε, που προκύπτουν στις διάφορες περιοχές. Βεβαίως ε, οι αρχές που μας διέπουν βασίζονται ε, στο βασικό κριτήριο της ε, από κοινού διαχείρισης. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερως που τα θέματα αυτά τα έχουμε περιλάβει στην ημερήσια διάταξη. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως το ελεγκτικό συνέδριο για την έκτακτη, για την ειδική μάλλον έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι υπέρ του Λίντερ. Και πάντα καλωσορίζω την πρωτοβουλία, της, τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτήν την ιδέα. Και κάθε δράση του. Αλλά έχω κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι όταν μιλάμε για το περιεχόμενο, τους στόχους ενός προγράμματος, είναι και οι στόχοι και το περιεχόμενο εξίσου σημαντικοί με το οικονομικό υπόβαθρο του προγράμματος. Με εκπλήσει λοιπόν το να λέει το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλό είναι το πρόγραμμα μεν αλλά η διαχείριση δημοσιονομική είναι κάπως προβληματική, υπάρχουν δυσκολίες εκεί κτλ. Όχι, η δημοσιονομική διαχείριση ενός προγράμματος είναι εξίσου σημαντικό κομμάτι ενός προγράμματος. Εάν υπάρχουν προβλήματα στη δημοσιονομική διαχείριση, τότε το πρόγραμμα δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Τότε είναι ένα κακό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε τις δύο αυτές πτυχές. Εγώ ε, καταγόμενος από χώρα στην οποία την εξουσία την είχαν επί δεκαετίες οι κομμουνιστές και εκείνοι προσδιορίζαν τους στόχους και μας έλεγαν είναι καταπληκτικοί οι στόχοι μας, έχουμε πολύ καλούς στόχους και προγράμματα, αλλά στην πράξη δυσκολευόμαστε λίγο και θα άρουμε τα προβλήματα στην εφαρμογή. Ε, μπορώ να σας πω ότι δεν ανέχουμε τέτοιου είδους δικαιολογίες. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς σε ένα πρόγραμμα λέει ότι είναι καλό πρόγραμμα αλλά έχει προβλήματα στην εφαρμογή, ε, το αποτέλεσμα για μένα είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα και άρα το πρόγραμμα είναι κακό πρόγραμμα. Και έτσι όπως είπα εξ αρχής, είμαι υπέρ του leader βλέπω ότι υπάρχουν πολύ κακά ε, πολύ κακές επιδόσεις ως προς την εφαρμογή, την υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν θεωρώ ε, καλό το να προκύψει το τέλος όλης αυτής της συζήτησης πως 10 χρόνια μετά ξαναδιαπιστώνουμε και άλλη μια φορά ότι υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει όμως. Πολλά από τα προβλήματα τα έχουμε διαπιστώσει εδώ και 10 χρόνια. Τα έχουμε εντοπίσει. Περάσανε 10 χρόνια χωρίς να αντιμετωπιστούν και έχουμε μπροστά μας ακόμη τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, εάν όλοι έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά, όπως μας δίνεται η εντύπωση εδώ, δεν θα έπρεπε να έχουμε τα ίδια προβλήματα 10 χρόνια μετά. Εφόσον εντοπίστηκαν πριν από 10 χρόνια τα προβλήματα αυτά, θα έπρεπε κάπως να έχουν αντιμετωπιστεί. Δεν γίνεται επομένως, δεν στέκει να λέμε ότι ο καθένας έχει κάνει τη δουλειά του σωστά. Και δεν λέω ότι πρέπει να δακτυλοδείξουμε κάποιους υπετίους, αλλά πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν έχει γίνει σωστά η δουλειά. Και συμφωνώ με τις προτάσεις του Ντέρεκ για να προχωρήσω σε κάποιες συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις για τις λεπτομέρειες. είναι ε, μερικές φορές πρόβλημα όπως επισημάνθηκε το γεγονός ότι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση των ε, σχεδίων ε, βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτή ήταν η παρατήρηση και από το ελεκτικό συνέδριο και την υποστηρίζω. Όταν για τα LAGs, για τις τοπικές ομάδες δράσεως έχουμε τέτοιου είδου ανάληψη της ευθύνης για την απόφαση, νομίζω ότι εάν δεν απατώμε και πιστεύω ότι πράγματι δεν απατώμε, εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με την πολιτική συνοχής συνολικά με την παραβίαση κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χαράσονται αυτές οι πολιτικές, με τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα διάφορα σχέδια και ως εκ τούτου παραβιάζεται η βασική αρχή της διαφάνειας στην πολιτική συνοχής. Γιατί αυτή την διαφάνεια την ορίζουν κάποιοι κανόνες, κάποιες διατάξεις. Αυτές οι διατάξεις υπαγορεύουν ποιος δημοσιεύει τι, πότε. Και δεν δέχομαι να υπάρχουν ε, οι ίδιοι κανόνες και σε κάποιους τομείς να παραβιάζονται, όχι απλώς να παραγνωρίζονται, αλλά να παραβιάζονται κατάφορα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τη διαφάνεια των στοιχείων. Και πρέπει να μπορεί κανείς να διαπιστώσει ξεκάθαρα ποια ομάδα, τοπική, τοπική ομάδα δράσεως έλαβε ποια απόφαση, σε τι αποτέλεσμα οδήγησε αυτή η απόφαση και τι χρησιμότητα είχε το αποτέλεσμα αυτό. Για τα προγράμματα Λίτερ, για το πρόγραμμα Λίτερ μάλλον και τα σχέδιά του, δεν βλέπουμε να ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση να ανατραπεί αυτή η πρακτική. Πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές διαφάνειας παντού. Και κάθε απόφαση για λόγους διαφάνειας ακριβώς πρέπει να καταγράφεται επακριβώς για κάθε απόφαση η διαδικασία με την οποία ελήφθη. Τώρα για τη σύσταση ε, του, συνεδρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα ήταν ε, κοντόφερμοι και άκαμπτοι οι κανόνες οι οποίοι θα μας οδηγούσαν να τις εφαρμόσουμε όπως έχουν χωρίς να λάβουμε υπόψη τις ε, πρακτικές και την λειτουργία των προγραμμάτων και πάνω απ' όλα τη μεταρρύθμιση των πρακτικών αυτών. Όταν έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα αυτή της ε, λήψης των αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο που επεσήμανε και ο εισηγητής, νομίζω ότι πρέπει να ε, δούμε ότι όταν έχει ληφθεί μία απόφαση δεν θα πρέπει να εμπλέκονται άλλες πηγές και θα πρέπει η τοπική διάσταση να λειτουργεί κατά τρόπον εμπλουτιστικό στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Πολλά είναι τα παραδείγματα βάσει των οποίων πιστεύω μπορούμε να διαπιστώσουμε πως έχει παρερμηνευθεί μερικές φορές αυτή η αρχή και όπου χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Άρα, κατά βάση, μπορώ να πω ότι οι τέσσερις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου είναι για μένα ικανοποιητικές, τις υποστηρίζω, είναι σημαντικές και στις συγκρούσεις συμφερόντων πιστεύω θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί από αυτό που προτείνει το συνέδριο. Στα δε ενεξελίξη σχέδια θα πρέπει πιστεύω να λάβουμε υπόψη και την αρχή της ευελιξίας που σύστησε ο Ντέρεκ Βόν. Από την άλλη πρέπει πάντοτε να ισχύουν οι κανόνες που έχουμε και στην πολιτική της συνοχής ε, και για την ανάπτυξη πέθρου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίλτερ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Ανέκαθεν θεωρούσα το Λίντερ πολύ δημοφιλές πρόγραμμα και με έκπληξή μου άκουσα ότι πολλές φορές κατά την προετοιμασία κάθε προγράμματος διαπιστώνεται σύγκρουση συμφερόντων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι έχουμε χρόνο, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα λάθη του παρελθόντος για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αναρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Όντως το Leader είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα. Όμως ο συνολικός προϋπολογισμός του αφορά σε σχετικώς μικρά ποσά. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς ε, τι γίνεται με το κόστος της διοίκησης για την προετοιμασία όλων αυτών. Τι κόστος συνεπάγεται ε, η διαχείριση της υποβολής των προτάσεων και πόσο είναι το κόστος τελικά που απολαμβάνουν οι τελικοί δικαιούχοι. Ε, κυρία Τσέσκοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, ίσως είναι αργά πλέον να ασκούμε κριτική, βλέποντας ότι το πρόγραμμα αυτό υπάρχει πάνω από μια δεκαετία τώρα και ενώ το έχουμε πάνω από δέκα χρόνια τώρα ε, έρχονται συστάσεις με τις οποίες βεβαίως συμφωνούμε. Δεν θα έπρεπε όμως να επικρίνουμε ε, τα τεκτενόμενα έστω και ελάχιστα. Εγώ θα ήθελα να το κάνω γιατί ε, η εμπειρία μου από την Τσεχία δείχνει ότι το διοικητικό άχθος είναι τεράστιο για τους δικαιούχους ε, σε σχέση και με όλες τις άλλες πρωτοβουλίες και τα ε, κονδύλια και γι' αυτό με εξέπληξε η έκθεση αυτή. Εάν δραματικά επιθυμούμε την απλούστευση, τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδεχομένως τα κονδύλια θα, θα, είχαν, θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει σε ανθρώπους που δεν χρειάστηκε να τηρήσουν ε, πρακτικά των πεπραγμένων στις συσκέψεις τους ή που θα μπορούσαν κάλλιστα να μοιράσουν τα κονδύλια, να τα μοιραστούν μεταξύ τους. Δεν χρειάστηκε να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ε, δεν χρειαζόταν ε, καθόλου δημοσίευση ε, της ενημέρωσης για το ποια προγράμματα επελέγησαν ή όχι. Δηλαδή, πολύ συχνά δεν υιοθετήθηκε αυτό το κριτήριο της ε, μη σύγκρουσης συμφερόντων και δεν υπήρξε καμία απέτηση για διαφάνεια. Και η διαφάνεια είναι μια λέξη κλειδί που επαναλαμβάνουμε συνεχώς στην Επιτροπή μας και είναι η βασική απέτηση που θα, με την οποία θα πρέπει να πληρούν όσοι λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και όσοι ασχολούνται ε, με την, ε, με την κατανομή των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλω δηλαδή να πω ότι εξεπλάγει σφόδρα διότι είδα ότι παραμένουν κάποια λεπτά ζητήματα και περιπτώσεις στις οποίες κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν είχε εφαρμοστεί σε άλλα προγράμματα. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο τελικός δικαιούχος είναι εξαιρετικά επαχθείς, δηλαδή είναι δύσκολο να τις ε, ε τηρήσει ε, κανείς από πλευράς ε, διοικητικής. Βεβαίως είναι καλό το ότι η Επιτροπή μας ασχολείται με αυτό το θέμα και πρέπει να εκφράσουμε τη συμφωνία μας με τις συστάσεις έστω και αν ήρθαν αργά. Θα έπρεπε όμως οι συστάσεις αυτές και οι έλεγχοι αυτοί να είχαν ε, προκύψει νωρίτερα. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ για το προσελεκτικό συνέδριο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Το πρόγραμμα αυτό, το Leader, το έχουμε εδώ και 20 χρόνια. Και η έκθεση είναι για μας καταστροφή. Καταστροφή πραγματικά. Δηλαδή, ερωτά κανείς τι να κάνουμε πια, πώς είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά χρήματα να τα χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, τη δήλωση του οικονομικού συμφέροντος του εμπλεκομένου. Βλέπουμε ότι δεν δίδεται σε μια τουλάχιστον ε, ομάδα δράση, τοπική ομάδα δράση που έχει ελεγχθεί. Δεν γίνεται δηλαδή σωστά η δουλειά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το leader το γνωρίζουμε όλοι. Και θέλουμε βεβαίω να συνεχιστεί και να λειτουργεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα αυτό. Να λειτουργεί όμω σωστά. Και δυστυχώ αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Δεν έχουν γίνει αρκετέ προσπάθειε. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιοριστούμε σε κάποια συμπεράσματα που θα λέγανε «Α, να διορθώσουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο κάποιες διορθωτικές κινήσεις». Είναι 20 χρόνια που υφίσταται το πρόγραμμα αυτό. Είναι δυνατόν να διατίθενται ευρωπαϊκά κονδύλια κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς κανέναν έλεγχο. Όχι, θα πρέπει να αλλάξουμε ριζικά, να διαρωτηθούμε αν πρέπει να επιφύσταται ακόμη το πρόγραμμα αυτό. Η Φερρυπίν βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν καταβληθεί κάποια ποσά για ε, πινακίδες οδικές. Είναι δυνατόν με χρήματα του Λίντερ να, πληρωθούν, να πληρωθεί η σήμανση στον δρόμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά μέτρα για αυτήν την υπόθεση και να δούμε στο μέλλον να τα αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει ο Σέλφος Βον να ολοκληρώσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αισθανόμαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για το επέδο και τον όγκο της συζήτησης αντιπαράθεσης που είχαμε στην υπόθεση αυτή. Νομίζω θα πρέπει, όπως είπε και ο κύριος Μιούλτερ, να εξετάσουμε το πόσο κοστίζει η διαχείριση. Όπως λέει και η έκθεση, από το 12% μέχρι το 2% ανέρχεται το σχετικό κόστος. Ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το κράτος δηλαδή. Επίσης ευχαριστώ και τον συνάδελφο κύριο Ντόιτ για τα σχόλιά του και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνει στην ε, ορθή λειτουργία του λίντερ. Πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε υπόψη ότι το leader έχει σημασία όσοι σημασία έχουν και τα σχέδια τα οποία προκύπτουν από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα το ίδιο αυτό καθένα αυτό, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε σχέδια αξιόλογα, σχέδια από τα οποία να υποφελείται και η τοπική κοινότητα, κοινωνία καλύτερα. Περιμένω επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτάσεις ε, για διαχείριση, καλύτερη διαχείριση στο μέλλον, τις οποίες ε, ασφαλώς και περιμένουμε με ε, αδημονία και πιστεύουμε θα είναι χρήσιμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Λαζάρου για την παρουσία του εδώ, για την ε, έκθεση που μα παρουσίασε. Πιστεύω ότι συμφωνούμε στα πάντα. Ένα-δύο σημεία ίσω ε, να εντοπίζουμε διαφωνίε, αλλά και πάλι και σε αυτά που υπάρχουν κάποιες διαφωνίες δεν απέχουμε πολύ μεταξύ μας. Πάνω απ' όλα επιβάλλεται η διαφάνεια πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα πρακτικά των εργασιών των τοπικών ομάδων δράσεως να δημοσιεύονται για να γνωρίζουμε τι κάνουν αυτές οι ομάδες δράσης. Οι δηλώσει οικονομικού συμφέροντος πρέπει πάντοτε να κατατίθενται και νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ του σημαντικού και του ασήμαντου ε, συμφέροντο ε, που επεσήμανε το συνέδριο ότι μερικέ φορέ δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η διάκριση και το δέχομαι αν μου το λέει το συνέδριο, αλλά ίσω θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σχετικέ προτάσει ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη σχετική διάκριση όταν υπάρχουν προβλήματα. Επίση, η περαιτέρω διαχείριση σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ένα άλλο ζήτημα, όπου έχουμε παραδείγματα νομίζω σχεδίων που αποδεικνύεται πως είναι πολύ επιτυχημένα και που θέλουμε να συνεχιστούν και να επεκταθούν. Φέρει την, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα την Ουαλία ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο είχε ξεκινήσει με την επέκταση της ευρυζωνικής ε, τεχνολογία στην περιοχή μα χρειάστηκε να επεκταθεί το σχέδιο αυτό, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του, χρειάστηκε να ληφθεί σχετική απόφαση. Εδώ νομίζω χρειάζεται κάποια ευελιξία και νομίζω ότι υπόθηκε από τον κύριο Λαζάρου ήδη πω ε, έχει προβλεφθεί, έχει εισαχθεί η ιδέα τη ευελιξία μέσα στο σύστημα, έτσι θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο για να είμαστε βέβαιοι ότι όταν είναι καλά τα σχέδια αυτά, όταν είναι bottom-up, όταν ξεκινάνε από τη βάση, όταν είναι ωφέλιμα για τι τοπικέ κοινωνίε θα πρέπει να τα διαφυλάτουμε, να τα προστατεύουμε και να επιτρέπουμε την ε, συνέχισή του. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία για όλα αυτά τα σχέδια. Τα σημεία, συγγνώμη. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Για πολύ λίγο, παρακαλώ, σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερως να εκφράσω την, ε, το σεβασμό ε, του ελεκτικού συνεδρίου στι ανησυχίε που εξέφρασε ο εισηγητή για τα σημεία 1 και 2 ιδιαίτερω. Βεβαίω θα συμφωνήσω ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί το ποσοστό επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα να τηρηθούν και οι βασικέ αρχέ που διέπουν του δημοσιονομικού κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ λέει ο Πρόεδρο. Περνάμε στο σημείο 9. Τη ημερήσιας διάταξη, ε, την ειδική έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου ελέγχη σχετική με την ζάχαρη. Ο κύριος Κυλακάκης έχει το λόγο παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, διότι μιλούμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στην κοινή γεωργική πολιτική μας, η οποία είχε να κάνει με διαρθρωτικά ταμεία και κονδύλια ύψους 6,2 δις ευρώ. Βασική στόχη της μεταρρύθμισης ήταν η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ζάχαρης, αλλά και η σταθερότητα των αγορών και ε, η διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας ζάχαρης, προμήθευσης με ζάχαρη της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε οικονομικά κίνητρα ώστε η παραγωγή ζάχαρης να τεθούν εκτός αγοράς. Σε γενικές γραμμές οι στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν στέφθηκαν με επιτυχία. Επιτεύχθηκε ο στόχος της αυξημένης ανταγωνιστικότητας και γεφύρωσης ε, της, ε, του χάσματος ε, της τιμής μεταξύ της Ευρώπης και του υπολείπου κόσμου. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες και όλοι ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από τις λεπτομέρειες. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει εκφράσει διάφορες επιφυλάξεις με τις οποίες δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Πρώτον, επιφύλαξη ως προς το, ε, το μέτρο της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται μόνο στις περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να εξετάσει την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε παραγωγού και δεν αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή για να συλλέξει στοιχεία από την ε, βιομηχανία ζάχαρης ή από τους παραγωγούς. Δηλαδή δεν έχουμε στοιχεία για το τι συνέβη ακριβώς επί τόπου. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για αυτό το θέμα. Τα στοιχεία για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χρήσιμα και δεν τα έχουμε αυτά, τα στερούμαστε. Θα μας ήταν χρήσιμα για να εξετάσουμε και όντως, αν όντω οι προσπάθειές μας ε, πέτυχαν επί τόπου, αλλά θα μας χρησιμεύαν και για την εξέταση ε, των μελλοντικών προοπτικών της κοινή γεωργικής πολιτικής. Για να μπω τώρα στις ε, λεπτομέρειες, θα ήθελα να θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, γιατί μεγάλη μεγάλη παραγωγή ζάχαρης που παρετήθηκαν από την ποσόστοσή τους, δεχόμενη τη μετατροπή και αξιοποιώντας τα ε, διαρθρωτικά ταμεία για να τεθούν εκτός αγοράς. Γιατί δεν μας έδωσαν στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια αυτά. Και το ρωτώ αυτό διότι όπως λέει και το ελεκτικό συνέδριο υπήρξαν παραγωγοί οι οποίοι έκλεισαν εργοστάσια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως άνοιξαν νέα εργοστάσια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πληρώσαμε χρήματα εμείς ως Ευρωπαίοι φορολογούμενοι για να επιχορηγήσουμε τη σύσταση και δημιουργία εργοστασίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θεμητό το ερώτημα πιστεύω. Ε, δεύτερο ερώτημα. Όσον αφορά τη βιομηχανία ζαχαρότευτλου. Ξέρετε ότι η παραγωγή ζαχαρόταυτλου που είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο έχουμε συμπεριλάβει την βιομηχανία, της ζάχαρης στην κοινή γεωργική πολιτική. Το λέω αυτό διότι δεν μπορεί κανείς να έχει παραγωγή ε, ζαχαρότευτλου χωρίς ε, ε, βιομηχανία ζάχαρης. Δηλαδή Υπάρχει σύνδεση, ένα κοινό πρόγραμμα γεωργίας και βιομηχανίας για την παραγωγή ζάχαρης από το τέφτλο. Ωστόσο, στα εργοστάσια ραφιναρίσματος δεν παράγεται ζάχαρη από ζαχαρότευτλο στην Ένωση. Αυτό είναι ένα προϊόν που προέρχεται από τροπικές χώρες. Μιλούμε δηλαδή για μια ε, βιομηχανική δραστηριότητα η οποία επηρεάζεται θετικά από την τιμή της ζάχαρης στο εσωτερικό της Ένωσης. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, γιατί έλαβαν ε, ενισχύσεις και πολλές ενισχύσεις, 50 εκατομμύρια ευρώ αν δεν απατώμε ε, με αυτή τη μεταρρύθμιση. Ποιο ήταν το δημόσιο αγαθό που εξυπηρετήθηκε με αυτά τα κονδύλια διότι ήταν κάτι που δεν ε, είχε συμπεριληφθεί στη μεταρρύθμιση αρχικά. Και ένα τρίτο ερώτημα που έχει να κάνει με την, με την ποσόστοση για την ισογλυκόζη, η οποία παράγεται από τον αραβόσιτο και άλλες πρώτες ύλες, ε, των οποίων οι τιμές δεν επηρεάστηκαν από τη μεταρρύθμιση ε, της κοινή οργάνωσης αγοράς ζάχαρης. Άρα, γιατί εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον με τις ενισχύσεις τους παραγωγούς ισογλυκόζης από τη στιγμή που η δική τους πρώτη ύλη δεν επλήγει, δεν άλλαξε η τιμή της με την μεταρρύθμιση στην αγορά της ζάχαρης. Και ένα τέταρτο ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον και το οποίο επισημαίνει και το ελεκτικό συνέδριο όντως έχει να κάνει με τα ωφέλη από τη μείωση της τιμής, ωφέλη τα οποία τελικά δεν απόλαυσε ο τελικός καταναλωτής. Και ε, ήταν ωφέλη που αφορούσαν τελικά, και αποδείχθηκε αυτό, ε, μόνο ε, στη βιομηχανία. Δηλαδή, μειώθηκε η τιμή, αλλά δεν την είδαμε εμείς, δεν την είδαν οι ψηφοφόροι μας, δεν την... Δεν είχαν πρόσβαση σε αυτοί οι καταναλωτές. Ερωτώ λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης αυτής, τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η μείωση της τιμής της ζάχαρης ε, χίδιν ε, θα περάσει τελικά, θα φτάσει μέχρι τον τελικό καταναλωτή ε, λιανικής. Και ένα τελευταίο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι η διαθεσιμότητα της ευρωπαϊκή ζάχαρης, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος ήταν 85% διαθεσιμότητα. Και όπως γνωρίζετε, η διαθεσιμότητα γεωργικών προϊόντων που παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής και κατοχυρώνεται από τη συνθήκη, τις συνθήκες. Ρωτώ λοιπόν, ε, αυτό το 85 είναι καλό ποσοστό, πώς το γνωρίζουμε αυτό, το ξέρουμε αυτό, θα μπορούσε να ήταν 90, θα μπορούσε να ήταν 80%. Δεν έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση για ή μάλλον δεν είδα η συζήτηση για τη διαθεσιμότητα να βασίζεται ε, σε σενάρια για τον αντίκτυπο της μη διαθεσιμότητας. Δηλαδή η συζήτηση δεν έχει βασιστεί σε εξέταση των διαφόρων ε, ενδεχομένων πιθανότητων. Ήταν μια συζήτηση ε, που έγινε στον αέρα, δεν βασίστηκε σε τεκμηριωμένα στοιχεία, δεν υπήρξε κάποια τεκμηρίωση, κάποια επιχειρηματολογία με βάση μελέτες συγκεκριμένες που να έχουν εκπονηθεί. Γιατί 85 και όχι 80 ή 90. Και θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Εξέτασα την ελληνική αγορά της ζάχαρης, η οποία επηρεάστηκε από αυτές τις μεταρρυθμίσεις αρκετά, γιατί... Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που χρειάστηκε να μειώσει στο μισό την ποσόστοση για τη ζάχαρη. Πέντε εργοστάσια είχαμε στην Ελλάδα, δύο έκλεισαν, ε, η ποσόστοση έπεσε στο ίμιση και είδα ότι τα υπόλοιπα τρία που υποτίθεται ότι η μεταρρύθμιση της ζάχαρης θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητά τους, αυτά τα τρία λοιπόν κινδυνεύουν να κλείσουν γιατί δεν παράγονται αρκετά τέφτλα ώστε να μπορούν να τα πάρουν τα εργοστάσια αυτά και να λειτουργήσουν στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο, στην ε, πιο αποδοτική ταχύτητά τους. Άρα είναι περίπτωση ε, στην οποία λέμε ότι η εγχείρηση πέτυχε αλλά δυστυχώς ο ασθενής απέθανε. Μήπως ισχύει αυτό τουλάχιστον σε ορισμένε περιοχές της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρετάν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολύ σύντομα θα μιλήσω Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον, τον εισηγητή σας για την εξαιρετικά επικοδομητική και αποδοτική ταυτόχρονα συνεργασία που είχαμε. Το έγγραφο εργασίας ε, το οποίο σας υποβάλλει σήμερα κατά την άποψή μου δίνει σαφέστατη παρουσίαση των κεντρικών μηνυμάτων αλλά και των συμπερασμάτων και των συστάσεων του συνεδρίου. Επομένως, αντί να επαναλάβω την έκθεση του κυρίου Σκυλακάκη, θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω κάποια σημεία. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος της μείωσης των 6 εκατομμυρίων τόνων ε, ε, όσον αφορά τις ποσοστώσεις ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτού του μέσου της, ε, του, του τέλους της υπερπαραγωγής και της πλεονοσματικής παραγωγής σακχάρεως, αυτός ο στόχος επετεύχθη. Όμως οι μειώσεις αυτές δεν αφορούσαν πάντα τα λιγότερο αποδοτικά εργοστάσια. Στην ουσία ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη-μέλη δεν είχαν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε σωστά να στοχεύσουν την μείωση ε, παραγωγικότητας. Ε, και επομένως 2,4 εκατομμύρια, δηλαδή 47% των 6 εκατομμυρίων, εγκατελείφθησαν από, ε, παραγωγής, από παραγωγούς ε, των οποίων ήταν ε, θεωρητικώς ανταγωνιστικά τα εργοστάσια κρίνοντας από τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο σημείο παράλληλα με την γενικότερη κινητροδότηση όσον αφορά την εγκατάλειψη των ποσοστώσεων, νέες ποσοστώσεις 1,5 εκατομμυρίων τόνων προσφέρθηκαν στις επιχειρήσεις. Αυτό το μέτρο μπορούσε να δικαιολογηθεί έτσι ώστε να υπάρξει ευελιξία στο σύστημα και για να επιτρέψει στις πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσα σε ένα δηλαδή ευρύτερο πλαίσιο μείωσης θα μπορούσαν κάποιες ανταγωνιστικές μονάδες να αυξήσουν την παραγωγή τους. Διαπίστωσε όμως το συνέδριο ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν επιτύχει ε, τις ε, ποσοστώσεις γρήγορα τις εγκατέλειψαν είτε ε, αφού τις αγόρασαν είτε αφού τους είχαν δοθεί. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν δόθηκαν και κατανεμήθηκαν σωστά αυτές οι ποσοστώσεις. Τέσσερο, τέταρτο σημείο. Η Ένωση από εξαγωγός έγινε εισαγωγός ακχάρεως. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον τρεις όμιλοι παραγωγής ακχάρεως που είχαν λάβει ε, βοηθήματα ε, για, το κλείσιμο εργοστασίων και ε, στην ευρωπαϊκή επικράτεια τελικά προχώρησαν την παραγωγή τους, την προώθησαν προς εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας. Αυτό στο μέλλον θα πρέπει να αποφευχθεί. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Και οποιαδήποτε κίνηση ενδεχομένως θα έχει κάποια επίπτωση στην παραγωγή ζάχαρης θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί από μέτρα παράλληλα τα οποία θα, ε, διασφαλίζουν την επάρκεια ζάχαρης που ήταν και ο αρχικός στόχος άλλωστε. Επόμενο σημείο. Η επίπτωση της μεταρρύθμισης στην τιμή της ζάχαρης όπως την πληρώνουν οι καταναλωτές. Το πεδίο είναι ε, ασαφές και δεν έχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση στη διάθεσή μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Σε γενικές γραμμές κατεδείχθη ότι η πραγματική μείωση της τιμής ζάχαρης χίδιν τελικά δεν μετακυλίστηκε στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές. Και επομένως, για να αντισταθμιστούν τα ασθενή σημεία της μεταρρύθμισης, το συνέδριο ε, κάνει μία σειρά ε, προτάσεων και συστάσεων που έχουν ενταχθεί στην έκθεση του εισηγητού σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Σκυλακάκη. Κύριε Κρετάν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για την ευκαιρία που μα δίνει να ανταλλάξουμε απόψει για τη μεταρρύθμιση τη ε, αγορά ε, ζάχαρη με βάση και τι συστάσει του Ελεκτικού Συνεδρίου και τι εκθέσει του κ. Σκυλακάκη. Και ιδιαίτερα, Πρόεδρε, δεδομένου ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης του 2006 ήταν μεγάλη επιτυχία. Οι θεσμικές τιμές περιορίστηκαν κατά 36% και η παραγωγή είναι πιο συγκεντρωμένοι στις περιοχές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ε, κερδοφορία. 78% αντί για 86% ε, επί του αντί για 68% ε, επί του ε, ποσοστού της ποσοστώσεως. Τώρα έχουμε μια, ένα καλύτερο προσανατολισμό, μια καλύτερη ευθυγράμμιση στην αγορά και κύριος στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η μείωση των τιμών και των διθρωτικών ταμείων που στήριζαν τους παραγωγούς, τον εγκατέλειπαν την παραγωγή ε, και την αντιστάθμιση των ε, δυσάρεστων για το περιβάλλον, των αρνητικών για το περιβάλλον ε, επιπτώσεων της μεταρρύθμισης. Και έτσι κάποιοι παραγωγοί παρατήθηκαν από τις ποσοστώσεις τους. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της ζάχαρης θα πρέπει να εξεταστεί και με υπόβαθρο τις γενικότερες ε, δεσμεύσεις και υποχρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς δηλαδή ε, δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρωτοβουλία τα πάντα πλην όπλων αλλά και την απόφαση της ε, ΠΟΕ σε σχέση με το καθεστώς τη ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου χάσαμε ένα πάνελ και εδώ, στην πρωτοβουλία χωρί όπλα, έχουμε ελεύθερη πρόσβαση για διάφορα προϊόντα στι αγορές Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένη και τη ζάχαρη και το πάνελ μίλησε για τον περιορισμό της επιδοτούμενης εξαγωγής ζάχαρης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόεδρε δεν είχε λύση άλλη από την απερικόψη της ποσοστός παραγωγής ζάχαρης προκειμένου να διαφυλάξει την απαραίτητη ισορροπία στην αγορά. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία που επισημαίνει το ελεκτικό ε, συνέδριο. Το κλείσιμο των 80 ε, εργοστησίων παραγωγής ζάχαρης η παραγωγή μειώνεται διαρκώ τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την μεταρρύθμιση της ζάχαρης. Κάθε μονάδα ε, αύξανε την παραγωγικότητά της ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας. Μέχρι το 2006 είχαμε 67 ε, κλεισίματα εργοστασίων από το 2000 στο 2006 με συνεχιζόμενη δηλαδή διαδικασία και η αναδιάρθρωση εξασφάλισε απλώς ένα ε, πλαίσιο νομικό, ένα μια βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να υποφεληθεί κανεί από το κλείσιμο των εργοστασίων, πράγμα το οποίο προηγουμένω δεν εξασφαλιζόταν. Επίση, η εξάρτηση από τι εισαγωγέ που αναφέρθηκε επίση. Η αύξηση εξάρτηση από εισαγωγέ δεν προκύπτει ω αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση στην αγορά τη Αχάρη. αλλά ω αποτέλεσμα των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω της πρωτοβουλία του 2001, τα πάντα πλην όπλων, που άνοιξε τις αγορές Ευρωπαϊκή Ένωση για εισαγωγέ από τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη του κόσμου. Και έτσι, πολλά από αυτά κράτη έχουν σημαντικό δυναμικό εξαγωγή σακχάριου. ελήφθη λοιπόν η πολιτική απόφαση να επιτραπεί στα κράτη αυτά να εξάγουν προ την κοινότητα. Η μεταρρύθμιση της Ακχάριος ε, επίσης αναφέρθηκε ως παράγον στη λήψη αυτής της απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, σε υποτιθέμενη περίπτωση υπό ελλειπούς κάλυψη των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε ε, ποσότητες ακχάρους που κανονικά θα εξάγονταν χωρίς επιδοτήσεις να τις εισαγάγουμε πολύ γρήγορα στην ποσόστοση. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ε, έλλειψη από την αγορά. Αναδιάρθρωση και επανεγκατάσταση και σχετική ενίσχυση. Η, επανεγκατάσταση έχει ενίσχυση στην επανεγκατάσταση έχει σαν στόχο ε, περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο μέλλον ένα εργοστάσιο να μπορεί να κλείσει και όχι μόνο το εργοστάσιο αλλά να δοθεί βοήθεια και για την αναδίπλωση του εργατικού δυναμικού, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών συνεπειών κτλ. Και θέλω εδώ πρόεδρε να υπογραμμίσω ότι είναι αμφίβολο το κατά πόσον προσπάθει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των ε, περιπτώσεων επανεγκατάστασης ε, των οικονομικών παραγόντων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να είναι συμβατές. Θα μπορούσε δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τρόπο συμβατό με του κανόνε του ΠΟΕ να παρεμποδίσει τέτοιου είδου μεταγκαταστάσει σε άλλα κράτη του κόσμου. Περιορισμοί δηλαδή σε επενδύσει θα ήταν πολύ δύσκολο να επιβληθούν νομότυπα. Και βέβαια αυτό θα σήμαινε ταυτόχρονα και ενίσχυση τη ανα... ενίσχυση για την αναδιάρθρωση. Ε, η μεταρρύθμιση λοιπόν συνέβαλε τα μάλα, αν και δεν ήταν μοναδικό παράγοντα, στην κάλυψη του κενού μεταξύ των ε, τιμών ε, των εσωτερικών με αυτών του εισαγόμενου προϊόντος ε, και έτσι έχουμε πολύ λιγότερου κινδύνους επανεγκατάσταση από ό,τι στο παρελθόν για τα δικά μα εργοστάσια. Και για να μιλήσω τώρα για τα σχόλια του κ. Σκυλακάκη. Καλωσορίζω βέβαια το γεγονό ότι ο κ. Σκυλακάκη αναγνωρίζει πω η μεταρρύθμιση στέφθη με επιτυχία, αυτό το πρώτο του σχόλιο, και έτσι τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου, μέσα στην εκθεσή του και τα λοιπά σχόλια και συστάσεις του κυρίου Σκυλακάκη, νομίζω μπαίνουν στην κατάλληλη προοπτική, με δεδομένο το ότι έχει στεφθεί με επιτυχία μεταρρύθμιση. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η βασική αρχή τη μεταρρύθμισης ήταν την τελική απόφαση για την διατήρηση, του περιορισμού ή την εγκατάλειψη ακόμα της παραγωγής, να την επαφίουμε στην απόφαση της ίδιας της επιχείρησης παραγωγής ή επεξεργασίας σακχάρους, με βάση και τις τιμές της αγοράς. Οι ίδιες λοιπόν επιχειρήσεις θα πρέπει με βάση οικονομικά στοιχεία οικονομική αξιολόγηση της κατάστασης να αποφασίζουν σε ποιο βαθμό είναι σε θέση να επιβιώσουν σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, εκεί δηλαδή όπου οι τιμές μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη και κατά 36%. Ε, οι επιχειρήσεις θα πρέπει μόνες τους να αποφασίσουν εάν θέλουν να αξιοποιήσουν το ε, Ταμείο Αναδιάρθρωσης και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο το να προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια ε, εργοστάσια επεξεργασίας ζάχαρη είναι ε, παραγωγικά και ποια δεν είναι ή μάλλον αποδοτικά. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουν οι επιχειρήσει μόνο του. Και ο κύριο Κυλακάκη, άλλωστε στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην περίπτωση του ελληνικού εργοστασίου, των ελληνικών εργοστασίων Σακχάριο, τα οποία επίση εκλήθησαν να λάβουν τι αποφάσει του, να κάνουν την αξιολόγηση του κατά πόσο θα μπορούσαν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον τη αγορά ζάχαρη και αν δεν είναι επιτυχία αυτή τη στιγμή, μπορεί στο μέλλον να είναι πιο αποδοτικά αυτή τη στιγμή που έχει υψηλή ε, τιμή η ζάχαρη, ίσω ε, να έχουν κάποιε πιθανότητε. Αλλά εάν δεν διαφυλαχθούν αυτέ οι τιμέ, μπορεί η οικονομική του αξιολόγηση να μην ήταν και πολύ σωστή. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας ζάχαρης νομίζω είναι αμφισβήτητη. Η παραγωγή της ζάχαρης αυτή τη στιγμή δρούν μέσα σε, μια, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό με χαμηλότερες θεσμικές τιμές και με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. η μεταβατική ενίσχυση για την ε, επεξεργασία ε, που παράγει το 72% της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει σημαντική συμβολή στην αγορά ε, ζάχαρης και γενικότερα τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταβατική λοιπόν αυτή ενίσχυση σημαίνει για τα εργοστάσια αυτά επεξεργασία ζάχαρης ότι μπορούν να προσαρμοστούν ε, στις νέες συνθήκες αγοράς και μάλιστα στις χαμηλότερες τιμέ. και έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια, η σταθερότητα στο μέλλον της αγοράς ζάχαρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσθετη ποσόστοση ισογλυκόζες Η ισογλυκόζη παράγεται από σιτηρά κυρίως και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως υποκατάστατο σάχαρης. Ως αποτέλεσμα αυτής της ε, μεταρρύθμισης μπορούν οι παραγωγοί ζαχαρής να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες τιμές των τεύτλων και έτσι να εξισορροπήσουν τη διαφορά τιμές σε σχέση με τους παραγωγούς ισογλυκώσεις. Και εδώ η ισογλυκώση έχει πρόσθετες ε, ποσοστώσεις, πράγμα που της επιτρέπει να ε, εκμεταλλευτεί της οικονομίας κλίμακος. Διαφορετικά, η σογλυκόζη θα είχε χαθεί από την ευρωπαϊκή αγορά και βέβαια η κατανάλωση σιτηρών θα είχε σημαντικά μειωθεί, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί ε, στόχο μας και δεν είναι προς το συμφέρον μας. Όσον αφορά τις τιμές καταναλωτού, ακριβώς στη συνέχεια της μεταρρύθμισης του 2006 θεσπίστηκε ένα σύστημα παρακολούθησης των τιμών καταναλωτού για να εξασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, ένα σύστημα το οποίο επιβεβαιώνει πως εν γέννη τιμές αγοράς ακολουθούν τη μείωση των θεσμικών τιμών που προσδιορίσε η μεταρρύθμιση και η Επιτροπή έχει αναλάβει και μια έκθεση για την εξέταση της ε, πορείας της τιμής άχαρης, για να δώσουμε επιστροφό στην υπόθεση αυτή. Και μετά την αξιολόγηση ε, της πολιτικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια εκ των υστέρων αναθεώρηση, επισκόπηση των μέτρων ε, μετά την ΚΑΠ που αφορούν τη ζάχαρη. Επίσης, Πρόεδρε, η μεταρρύθμιση αυτή έχει ξεκινήσει το 2006 και έχει εφαρμοστεί διαφορετικά στάδια. Κάποια από τα σχετικά μέτρα που έχουν να κάνουν και με τα ε, μέτρα αντιμετωπίσης απερίμωσης ξεκίνησε το 2007 μόνο. Ε, μόνο τώρα βλέπουμε την ουσιαστική αποτελεσματικότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων και με υπόβαθρο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξετάσει στην αξιολόγηση των μέτρων της ΚΑΠ που εφαρμόζεται το τομέα της ζάχαρης και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Η αξιολόγηση αυτή θα αρχίσει όπως προβλέπετε το Δεκέμβριο. Τώρα δηλαδή. Αποτελέσματα περιμένουμε μέχρι τα τέλη του 2011. Και φαντάζομαι πρόεδρε με αυτά που είπα απάντησα επαρκώς στις παρατηρήσεις του κυρίου Κρετάν, του κυρίου Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κυλακάκης για τα τελικά συμπεράσματα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, λεπτομερείς απαντήσεις που έδωσε σε όλα τα σημεία τα οποία είχα θίξει εγώ. Παρ' όλα αυτά εξακολουθώ να έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ε, η μία επιφύλαξη είναι η εξής. Βεβαίως ε, δεν θέλαμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουν οι ε, παραγωγοί της ε, ε, ζάχαρης με τα χρήματα, αλλά γιατί να μην έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Ένα πράγμα είναι ότι δεν αποφασίζουμε, δεν εμπλεκόμεθα στην απόφασή τους, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα διαφάνειας. Γιατί αυτό που ανέφερα και εγώ, αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο, για μονάδες εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας ε, δεν αναφέρεται στο ότι δεν έχουν δικαίωμα να ε, χτίσουν εργοστάσια εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας ε, αλλά ότι ευρωπαϊκά χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την οικοδόμηση και την οργάνωση αυτών των μονάδων. Εκεί είναι το ζήτημα και έγκυται στη διαφάνεια. Ισογλυκόζη και ζαχαροκάλαμο. τελικά θέλουμε να κρατήσουμε στη ζωή τις, ε, τα, ε, τις ραφινερίες ε, της ζάχαρης με, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λειτουργούν όμως με εισαγόμενα ζαχαροκάλαμα και από την άλλη πλευρά γιατί τότε δεν βοηθάμε και τους ε, παραγωγούς ε, ε, ζαχαρότευτλων γιατί κάθε φορά που κλείνει ένα εργοστάσιο ζάχαρης χάνουμε και ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών ζαχαροτεύτλων. Επομένως δεν είναι δυνατόν να δίνουμε μονάχα χρήματα για το ζαχαροκάλαμο και από την άλλη μεριά να κλείνουν μονάδες. Τώρα για την ισογλυκόζη δεν έχω οικονομικά στοιχεία και δεν γνωρίζω κανένα, καμία οικονομική αρχή που να αναφέρεται στην ίση μεταχείριση, equal treatment, χωρίς να ξέρουμε όμως, να έχουμε ορίσει εκ των προτέρων, τι σημαίνει αυτή η μεταχείριση, ποιο είναι το treatment. Για να τελειώσω, να πω το εξής. Είναι σημαντικό να βλέπουμε την μεταρρύθμιση όχι μονάχα στα επιτυχή της σημεία αλλά και στα ασθενέστερα σημεία και είναι καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ιδιαίτερο τα ασθενή σημεία αυτής της ε, μεταρρύθμισης και θα είναι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου 8 2010 «Βελτίωση της επίδοσης των μεταφορών στους διευρωπαϊκούς σιδηροδρομικούς άξονες». Ερώτηση. Αποδείχθηκαν άραγε αποτελεσματικέ οι επενδύσει στι σιδηροδρομικές υποδομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνάδελφο Μπαλτσίτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας προτείνω να δώσουμε το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας να μιλήσει πρώτα για το πρώτο το ελεκτικό συνέδριο και μετά εγώ. Ευχαριστώ, ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω μια έκθεση η οποία αφορά κατά κύριο λόγο στην επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σιδηροδρομικών υποδομών και στόχος είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα. Αυτές οι επενδύσεις όντως βελτίωσαν τις επιδόσεις των μεταφορών στα διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Το ελεκτικό συνέδριο για τη δουλειά του βασίστηκε ε, σε αυτό το οποίο είχε οριστεί το 2004 στους προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 19 σχετικά ε, προγράμματα και σχέδια ε, για τους σιδηροδρομικούς διευρωπαϊκούς άξονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγα συντόμως θα αναθεωρήσει αυτούς τους προσανατολισμούς. Ε, είναι ανάγκη να γίνονται επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές και οι επενδύσεις αυτές είναι πολύ υψηλές. 92 δις ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί σε σιδηροδρομικά σχέδια και έργα μέχρι το 2007 και βάσει εκτιμήσεων άλλα, δύο, ε, άλλα 200 δις ήταν απαραίτητα, χρειάστηκαν για να ολοκληρωθούν τα, έργα, τα μεγάλα αυτά έργα. Το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε λοιπόν την αποδοτικότητα βάσει 8 ε, σιδηροδρομικών αξώνων και είχαμε ένα δείγμα 21, 21 τομέων που είχαν συγχρηματοδοτηθεί. Το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε ε, τομείς που ανταποκρίνονται σε ευρωπαϊκές επενδύσεις 8,6 δις ευρώ μέχρι και το 2006. Εν συντομία, οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ε, σιδηροδρομικές υποδομές πράγματι αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και αποδοτικές. Αυτό το ε, έχει βεβαιώσει το ελεκτικό συνέδριο. Η Ένωση συνέβαλε στο άνοιγμα νέων προοπτικών ε, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή καταφατική είναι η απάντηση, ναι, τα μεγάλα έργα ε, σιδηροδρομικών υποδομών ε, που γίνονται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά οδήγησαν στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης, στην αύξηση της ε, χωρητικότητας, της αποδυτικότητας και άνοιξαν νέοι δρόμοι πολύ σημαντικοί. Πάντως, το ελεγκτικό συνέδριο επισήμανε επίσης και συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, να βελτιωθεί ο μηχανισμός σωστής στόχευσης των επενδύσεων της Ευρώπης, να υιοθετηθούν μέτρα επιπρόσθετα ε, ώστε να μειωθούν τα εμπόδια και η δισκαμψία που ενίοτε υπάρχει. Το μήνυμα του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι το εξή. Καλούμε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου ε, κατά την εξέταση των μεταρρυθμίσεων που θα γίνουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα ώστε να βελτιωθεί ε, ώστε τον περισσότερο η χρήση των πόρων της Ένωση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο κ. Μπάλτσιτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον ε, κύριο Γκράθρεν ιδιαίτερος για την πολύ καλή έκθεση. Ήταν πολύ σημαντικό ε, να είναι τόσο καλή έκθεση αυτή την πρώτη φορά. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα πως μέσω της συγχρηματοδότησης η ανάπτυξη των ε, υποδομών επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων μεταφορών, δρομικό μεταφορών. Ε, προβλήματα όμως τα οποία θα πρέπει πιστεύουμε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να ε, ρυθμιστούν τα προβλήματα αυτά δεν επισημένονται και θα πρέπει να δούμε καταρχά ποιο είναι οι κύριοι στριοδρομικοί άξονε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα ε, σχέδια προτεραιότητας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσθεμένη έξι της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε τους ορισμού, ώστε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και συγκέντρωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας με τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδορίσουν τα ε, σχέδια τα οποία έχουν προτεραιότητα με ε, γνώμονα την αποδεδειγμένη χρησιμότητα ή τις ανάγκες για το μέλλον σε ευρωπαϊκούς άξονες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό των σχεδίων ε, που είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση προσδιορίζουν μόνο ε, τις αναγκές με βάση το υφιστάμενο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν συμβουλεύονται δηλαδή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και όταν έχουμε να κάνουμε ιδιαίτερα δύσκολε γεωγραφικέ συνθήκε ή ιδιαίτερε ε, ανάγκε προστασία του περιβάλλοντο, αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και το κόστος αλλά και τη διάρκεια υλοποίησης των ε, σχεδίων. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη πριν από την έγκριση της χρηματοδότησης. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν υπόψη τους και τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών στην υπόθεση αυτή. Βελτίωση επίσης ως προς την κυκλοφορία των ε, τρένων υψηλής ταχύτητας έχει σημειωθεί. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτό να προχωρήσει και για, το, για τη μεταφορά φορτίου, αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας και σήματα διαφορετικά και ενοποίηση των πολλών διαφορετικών σιδηροδρομικών συστημάτων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη πολύ στενά για να τα βοηθήσει να περιορίσουν αυτά τα προβλήματα ασυμβατότητας. Επίσης πιστεύουμε ότι η εκτελεστική υπηρεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για να μπορεί να παρακολουθεί και την υλοποίηση των σχεδίων. Υπάρχουν κάποια θετικά πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Όταν ορίστηκαν δηλαδή οι συντονιστές των σχεδίων TNT, των ευρωπαϊκών δικτύων δηλαδή, βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα και οι επενδύσεις και αυτό αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα πίεσης για να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η λειτουργία των ε, σχεδίων προτεραιότητας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ορίζει τους συντονιστές ε, για εκείνα τα σχέδια τα οποία παρουσιάζουν τρεις δυσκολίες. Η ε, χρηματοδότηση επίσης των διασυνοριακών σημείων από τα οποία παίρνουν αυτά τα σχέδια των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να βελτιωθεί. Προσδιορίζονται συντονιστέ για τι διευρωπαϊκέ εκείνε που αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικέ, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί ε, η ποιότητα τη μεταφορά, κυρίω σε περιοχέ δύσβατε. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών να λάβει υπόψη τα εκρεμή και σημαντικά ζητήματα, να αναθεωρήσει δηλαδή με βάση τις μελλοντικές προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας, 15 σημεία τα οποία πιστεύω στο μέλλον θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε την κατάσταση σε περισσότερο βάθος. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για αυτή την ε, σε βάθος ανάλυση που έκανε, αλλά και για τη δουλειά όλη που έχει κάνει, παρά τις ε, ε, μετεωρολογικές συνθήκες όπως βλέπουμε από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την έκθεση. Ε, σε γενικές γραμμές είναι θετικό το ελεγκτικό συνέδριο ως προς τη συγχρηματοδότηση και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και θα δώσει και συνέχεια σε όλα αυτά όπως ε, Κάναμε και με την έκθεση του 2003 και του 2005. Ε, όλα αυτά εντάσσονται και στις πολιετής αποφάσεις στη συγκέντρωση των κονδυλίων, στον ορισμό των συντονιστών, αλλά και στο εργαλείο Jaspers της Γενικής Διεύθυνσης ε, για τις Περιφέρειες, βάσει της γνωμοδότησης των επιρρογνωμόνων. Ως προς τις συγκεκριμένες συστάσεις που διατυπώνει το ελεκτικό συνέδριο, ήδη εμείς έχουμε αναλάβει δράση από τότε που συζητήθηκε και καταρτίστηκε η έκθεση αυτή το 2008 και το 2009 και μπορώ να σας αναφέρω επιγραμματικά και τις δράσεις που έχουμε αναλάβει ε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και που θα συνεχίσουμε βέβαια και τα επόμενα. Καταρχάς ε, ζητήθηκε το δίκτυο για, τα διευρωπαϊκά δίκτυα να βασιστεί περισσότερο στα στοιχεία με, που έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Έχουμε φτιάξει μια τεχνική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα, ε, τους 6.600 τομείς των ευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία λεπτομερή για όλα τα χαρακτηριστικά ε, αυτό έχει γίνει από το 2007 και μετά, ώστε ε, να λάβουμε υπόψη μας τη συγκεκριμένη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, δουλεύουμε επίσης πάνω στο ρόλο των συντονιστών. Έχουν οριστεί τρεις ακόμα συντονιστές, κύριοι Βελάξ, Κόξ και Σαβαρή, για να ενισχυθεί ο ρόλος γενικά του συντονιστή και εν ώψη της αναθεώρησης, της επικείμενης αναθεώρησης, θα λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σας ώστε η προσέγγιση μας να έχει να κάνει με τον πυρήνα του δικτύου και να μην είναι αποσπασματική και κατακαιρματισμένη. Συμφωνώ και με την παρατήρηση που κάνατε ότι το δίκτυο είναι καταρκεματισμένο χρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση. Έχουμε διάφορους διαδρόμους, είτε για τις εμπορευματικές μεταφορές, είτε για άλλες. Και όλα αυτά θα τα εντάξουμε στις προτάσεις που θα παρουσιάσουμε το 2011. Τώρα, και το Jaspers, αλλά και η εκτελεστική υπηρεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TEN-T, ε, είναι ενεργά όργανα, επάνω από 200 άνθρωποι εργάζονται ε, πάνω σε αυτό το θέμα και με τις δημοσιονομικές προοπτικές θα έχουμε αποτελέσματα. Το 2008 ε, έγινε ένα, συστήθηκε μια ομάδα που ασχολήθηκε κυρίως με την ανταλλαγή απόψεων και την, ε, σε βάθος γνώση της κατάστασης. Το 2009 στην Ολλανδία, στη συνέχεια στην Πορτογαλία. Πολλά έργα ε, συγχρηματοδοτήθηκαν και πολλοί συμμετέχοντες κλήθηκαν να παραστούν σε αυτά τα εργαστήρια που οργανώθηκαν στην Ολλανδία, Πορτογαλία και αλλού και δύο φορές ετησίως υποβάλλονται ε, αυτές οι εκθέσεις που μας βοηθούν στην αξιολόγηση των μεγάλων έργων ώστε να προχωρήσουν. Τώρα, ως προς τους ε, κανόνες λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των ε, ευρωπαϊκών διαδρόμων. Σήμερα, σε ορισμένους ε, διαδρόμους αλλάζει το καθεστώς ή ε, τα έγγραφα δεν έχουν την ίδια μορφή παντού διαλειτουργικότητα, δηλαδή ε, είναι κάτι που υστερεί, υστερούμε σε αυτό, πρέπει να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Και το προσπαθούμε. Έχουμε υιοθετήσει το TSI, που είναι τα στάνταρ διαλειτουργικότητας για τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας, αλλά και για τους συμβατικούς σιδηροδρόμους. Βεβαίως πρέπει να εναρμονίσουμε ακόμα περισσότερο ε, την κατάσταση και στην επόμενη αναθεώρηση θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτές ακριβώς τις πτυχές. Η εναρμόνιση είναι δύσκολη ενίοτε ε, με την προσέγγιση που έχει να κάνει με τον πυρήνα του δικτύου. Ε, πιστεύω όμως τον Ιούνιο, τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς θα έχουμε πολύ ε, σημαντικές προτάσεις. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου έρχεται σε μια πολύ καλή χρονική συγκυρία. Μπορούμε να την αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να καταρτήσουμε καλύτερα προτάσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς. Στις προτάσεις θα λάβουμε απολύτως υπόψη μας τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ η συνάδελφος κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, τον κύριο Μπαλτσίτης, για αυτή την πρόταση εργασίας που μας έχει υποβάλει και για την έκθεσή του, η οποία περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα ε, στοιχεία που μας βοηθούν στη συζήτηση για τις μελλοντικέ προοπτικές των σιδηροδρόμων. Εγώ ασχολούμαι με τα θέματα αυτά στην Επιτροπή των Μεταφορών και θα ήθελα σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Και το λέω αυτό διότι με εκπλήσει, να το πω έτσι, ε, το περιεχόμενο ορισμένων συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου, ε, το οποίο ελεκτικό συνέδριο βεβαίως στοχεύει πάντοτε στη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά ε, κάνει συστάσεις πολιτικής χρειάς θα έλεγα το ελεγκτικό συνέδριο και ίσως έτσι παραγνωρίζει την ιστορική διαδρομή των, ευρωπαϊκών, ε, των διευρωπαϊκών δικτύων αν δεν υπολείπεται ως προς την ε, τις απαραίτητες γνώσεις και τα απαραίτητα στοιχεία πληροφόρησης που θα έπρεπε να έχει. Γίνεται μια πρώτη σύσταση η οποία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη υπομονή. Εμείς όμως ως Κοινοβούλιο έχουμε λιγότερο, λιγότερη υπομονή. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους οργανισμούς σιδηροδρόμων, τους εθνικούς, οι οποίοι εθνικοί σιδηρόδρομοι είναι αυτοί που αποτελούν και αποτελούσαν πάντοτε τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την διεύρυνση αυτού του διευρωπαϊκού χαρακτήρα των δικτύων. Δεν θα πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας τον στόχο μας, να μην παρεκκλίνουμε από την πορεία μας. Ε, ε, καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ξεπεράσει τα εθνικιστικά, αν θέλετε, πατερναλιστικά συμφέροντα, τα κρατικά συμφέροντα των κατατόπους εθνικών ε, σιδηροδρομικών οργανισμών οι οποίοι ε, πολύ συχνά δεν διασφαλίζουν την ε, διασωνοριακότητα και οι οποίοι πολύ συχνά εμποδίζουν και έχουν εμποδίσει αυτό τον ευρωπαϊκό κοινό σιδηροδρομικό χώρο τον οποίο εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά από τόσα χρόνια επιτέλους. Τώρα, ως προς τους συντονιστές, είναι αληθές αυτό που λέγεται. Θέλουμε ως Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει το ρόλο των συντονιστών. Όμως σε όλη αυτή την πορεία έχουν υπάρξει περιπτώσεις και αυτό το οποίο αφορά εμένα με τα ισπανικά έργα, με τα έργα στην Ισπανία, ε, είναι το εξής. Ενίοτε χρειάστηκε να αλλάξουμε συντονιστή, παρόλο που ε, ουσιαστικά φάνηκε ότι δεν τον εκδιώξαμε, αλλά ότι τον αποχαιρετήσαμε με όλους τους επένους. Αλλά χρειάστηκε να τον αποχαιρετήσουμε με όλους τους επένους, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος και προκειμένου να διευκολυθούν σχέσεις με κράτη-μέλη ε, των οποίων οι προτεραιότητες δεν έχουν καθόλου να κάνουν με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους και την, ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα εν γέννη. Επομένως, ε, θα πρέπει να βελτιωθεί και η δουλειά των συντονιστών. Όχι μόνο να ενισχυθεί ο ρόλος τους. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν λέει επίσης ότι ο προϋπολογισμός είναι κατάφορα ανεπαρκής. Στα τέλη του 2010 έχουμε δαπανήσει άνω του 90% του συνόλου του προϋπολογισμού για όλα τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα. Γιατί δεν το λέει αυτό το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός. Θα ήθελα να το δω στην έκθεσή του. Από εκεί και πέρα, ε, καλώς ε, αποφαίνεται ε, για τη βελτίωση ε, των μεταφορών επιβατών αλλά και των εμπορευμάτων. Ωστόσο, στα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τη συγχρηματοδότηση, τη συνοχή και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, διότι δεν μπορεί να γίνει συγχρηματοδότηση του ίδιου κομματιού τη διαδρομή, μπορεί όμω να υπάρξει αλληλοσυμπλήρωση. Αυτό δεν το σχολιάζουν καθόλου, ενώ θα μπορούσε να ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Και τέλο, κάτι το οποίο ε, αφορά εμένα προσωπικά και το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά, θα ήθελα το ελεκτικό συνέδριο να διερευνήσει περισσότερο την κατάσταση. Ε, αναφέρομαι βεβαίως στη γραμμή που μας συνδέει με τη Γαλλία. Και στην Ισπανία έχουμε πρόβλημα, ενώ μας, μας λένε ότι το κομμάτι της Γαλλίας δεν έχει πρόβλημα. Ισχύει αυτό. Επί Φράγκο ε, πάντοτε υπήρχε αυτός ο φόβος, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής εισβολής ε, η οποία θα περνούσε από τα Πυρηναία και θα έφτανε σε εμάς. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και χρειάζεται ένας τρίτος δρόμος. Το λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Και επιτέλους στις 18 Δεκεμβρίου θα περάσει τα σύνορα η πρώτη πομπή οχημάτων. Όμως από τη γαλλική πλευρά των συνόρων δεν έχει γίνει επαλήθευση της ηλεκτροδότησης του δικτύου. Επομένως, γιατί υπολείπονται εκεί, γιατί δεν έχουν κάνει τα μέλη. Δηλαδή θα περάσουν πλέον τα ισπανικά σύνορα από την Ισπανία προς τη Γαλλία, η πρώτη πομπή θα, την, θα τα περάσει, αλλά δεν έχουν οι Γάλλοι από την πλευρά τους ελέγξει την ηλεκτροδότηση. Γιατί. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έγραφο εργασία. Είναι πληρέστατο πιστεύω. και παρουσιάζει τις πιο σημαντικές πτυχές της εκθέσεως του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αυτό λοιπόν στις δρομικές μεταφορές δεν είναι τόσο ευρωπαϊκές όπως τα θέλαμε. Είναι πολύ έντονος ο παράγοντας, ο εθνικός ακόμη. Ενώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τίνουμε προς μία ε, ευρωπαϊκή τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Μεταφορών. Η κρίση με, τις, με την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία απέδειξε ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Και πιστεύω και ελπίζω ότι έχει και το ελεκτικό συνέδριο και ο εισηγητή παρουσιάσει πολύ σημαντικέ πτυχέ τη υπόθεση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά προγράμματα, Φερρυπίν, σύζευξη των Βαλκανικών κρατών ten ε, οι μεταφορές των ε, φορτίων. Ο συντονισμός των προγραμμάτων μεταξύ τους, οι προτεραιότητες που προσδιορίζονται, ώστε να έχουμε στο δυνατόν πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η έννοια του συντονισμού για μένα είναι μια καλή ιδέα, ναι, θα πρέπει να προσδοριστούν νέοι στον στο μέλλον. Ε, ωστόσο, σχέδια τα οποία έχουν αντίστοιχη ε, διαμόρφωση αφορούν τα ίδια κράτη-μέλη, καλό θα είναι να έχουν ίσως τον ίδιο συντονιστή για δύο διαφορετικά σχέδια. Το ελεγκτικό συνέδριο, μετά η Κομισιόν και μετά ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αντιδράσω ε, στα όσα είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ. Είναι προφανές ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι πολιτικό όργανο. Το συνέδριο εκλήθη να ε, αποφασίσει, να αποφανθεί επί της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Δεν είναι δικό μας θέμα να κάνουμε πολιτικές κρίσεις. Και όσο παλαιός Υπουργός Μεταφορών Βεβαίως θα μπορούσα να πω κι άλλα αλλά αυτά τα άλλα θα ξεπερνούσαν τις αρμοδιότητες ε, του ε, συνεδρίου. Και πρέπει να σας πω και ότι σας το αποκαλύπτω αυτό, ότι συχνά με σκουντάνε οι συναδελφοί μου και μου λένε «Δεν είσαι πια στην πολιτική θέση που ήσουν πριν», Τώρα είσαι στο ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω κυρία Ιάλα Σέντερ ότι θα μπορούσα να πω κι άλλα αλλά θα ξεπερνούσα σαφώς την εντολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους παρεμβαίνοντες σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ε, για τα θετικά σήματα τα οποία μας ενθαρρύνουν στη συνέχιση του έργου μας. Ευχαριστώ. η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση των σχολείων που διατυπώθηκαν, να πω στην κυρία Γιάλα Σέντερ ότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση για το μη άνοιγμα ε, των ε, ε, σιδηροδρόμων και έχει ξεκινήσει επιπλέον δράση ε, κατά των 14 αυτών χωρών. Ε, συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα ανοίγματο τη αγορά. Συμφωνώ με την κυρία Γιάλα Σέντερ. Δεν έχει γίνει άνοιγμα των αγορών ε, παρά την εφαρμογή της δέσμης των σιδηροδρόμων και όπως γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Γιάλα Σέντερ υπάρχει πρόταση για αναδιατύπωση της πρώτης σιδηροδρομικής δέσμης Όπως είπε όμως και ο κύριος Γκρετάν, δεν ε, αντιμετωπίσαμε αυτήν την ανάλυση, αυτό το θέμα. Στον κύριο Μαρινέσκου μπορώ να υπογραμμίσω την ε, επιθυμία μας όντως ε, για συνεργασία μεταξύ και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων οργανισμών, κυρίως όσον αφορά ε, τα κατά προτεραιότητα προγράμματα. Να σας πω ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες αυτές συγχρηματοδοτούνται ε, από τον προϋπολογισμό RTNT και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται αυτές τις διάφορες πρωτοβουλίες. Όμως και απαντώντας την ερώτησή σας, έχουμε ε, την πρόθεση να ε, συντονίσουμε τους, τις διάφορες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους συντονιστές και η κυρία Γιάλα Σέντερ και ο κύριος Μαρινέσκου έκαναν παρατηρήσεις σχετικά με τους συντονιστές. Είμαστε πεπισμένοι ότι ήταν σωστή η επιλογή. Οι συντονιστές κάνουν αναφορά ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μία φορά το χρόνο. Συμφωνώ βεβαίως ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και φυσικά οι συντονιστές πρέπει να πηγαίνουν επί τόπου έτσι ώστε να ε, καταδεικνύουν τα προβλήματα. Ε, όντως βγαίνοντας από το τούνελ Περπινιάν Φιγκέιρας ε, υπάρχουν ε, ε, σημεία των τροχιοδρομών με ηλεκτροδότηση 1,5 βόλτ και αυτό όντως δημιουργεί προβλήματα και θα πρέπει να τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά. γιατί όπως λέει και το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να συγκεντρώνουμε τόσα χρήματα για την οικοδόμηση ενός ε, διασυνοριακού τούνελ ε, και τελικά να ε, μην προχωράμε ένα πολύ μικρό κομμάτι του έργου το οποίο όμως θα είναι πολύ αποτελεσματικό για την σωστή ολοκλήρωση του έργου αυτού. Ο κύριος, ε, ε, ο συνάδελφος μάλλον, Μπάλτσιτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους και του Ελεκτικού Συνεδρίου και του, ε, της Επιτροπής για τα σχόλιά τους. Κατανοώ τις ανησυχίες που εξέφρασε η συνάδελφος Αγιάλα Σέντερ και βεβαίως ε, οι ανησυχίες αυτές ε, εντείνονται ε, και λόγω ιστορικών στοιχείων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι, σημαίνει, τι σήμαιναν σιδηρόδρομοι. Είχαμε και εμείς, ξέρετε, σιδηροδρόμους με την, στα σύνορα με τη Σοβιετική Ένωση την προηγούμενη δεκαετία έγιναν πολύ εντατικές συζητήσεις και εγώ σαν Υπουργός Μεταφορών επί τετραετία παρακολούθησα από κοντά τα θέματα αυτά. Βεβαίως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και ε, περιμένουμε με προσδοκία τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2011, κυρίως δε αυτές τις προτάσεις οι οποίες ε, θα καθορίσουν καλύτερα τους διευρωπαϊκούς άξονες. Η Ευρώπη χρειάζεται ε, μια ραχοκο... σιδηροδρομική ραχοκοκαλιά ή δύο τέτοιες σπονδυλικές στήλες σιδηροδρόμων είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να προχωρήσει σωστά ο σιδηρόδρομος. Ε, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ε, όλους όσους συμμετέσχουν στην συζήτηση και μακάρι οι σιδηρόδρομοι να γίνουν το κύριο μέσο μεταφοράς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που έμειναν παραπάνω από την ώρα τους. Όχι, όχι Πρόεδρε, με συγχωρείτε κυρία Χολμάιερ. Μια παράκληση. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση για το αίτημά μου να συζητήσουμε ε, την κατάσταση με το Ελεκτικό συνέδριο. Αν έχει δώσει κάποια απάντηση στο Ελεκτικό συνέδριο. Απάντηση. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Δεν αντελήφθη την ερώτηση. Το κοινοβούλιο, λέει η κυρία Χολμάιερ, Πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είχα ζητήσει από το Ελεκτικό Συνέδριο μέσω του Προέδρου Μπούζεκ να εξετάσει την ε, χρήση κονδυλίων και τους ελέγχους στο ΣΥΣ 2 μέσα σε μια ειδική έκθεση. Ε, ξέρουμε ότι έχει μια τέτοια επιστολή στο Ελεκτικό Συνέδριο. Τώρα βλέπουμε και πάλι αντιφατικά ποσά, ερωτώ εάν κάνει την επαλήθευση στο Ελεκτικού συνέδριο. Απάντηση. Το Ελεκτικό συνέδριο, πρόεδρε, εξετάζει τον τρόπο διάθεσης. Ε, δεν ξέρω αν αυτό θα ενταχθεί μέσα σε έκθεση ή σε επιστολή του Προέδρου μας προς το Κοινοβούλιο. Θα ενημερωθώ και θα σας πληροφορήσω. Πέρα στη συνεδρία